I think, dear colleagues, that we will start the meeting. And as you might remember, we have changed yesterday the agenda. Συνάδελφοι, αν θυμάστε, αλλάξαμε χτες την, ημερη, την ημερήσια διάταξη χτες ε, και αρχίζουμε με την έκθεση της κυρίας Μάνερ πρώτα και μετά θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες. Με τη σειρά που είχαν προβλεφθεί. Δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στη Ρίκα Μάνερ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις τροπολογίες τους. Λάβαμε αρκετές και χάρη σε αυτές μπορέσαμε να συντάξουμε αυτή την έκθεση και να αρχίσουμε τη σύνταξη συμβεβαστικών τροπολογιών με τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, υπάρχουν κάποια προβληματικά σημεία, αλλά πιστεύω και ελπίζω πως θα φτάσουμε σε συνένεση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κυριότερα σημεία. Βασική ανησυχία του Κοινοβουλίου είναι εξή, ότι δηλαδή σε αυτή την πρόταση κανονισμού για πρώτη φορά ο κανονισμός θα πρέπει να είναι αρκετά σαφής έτσι ώστε το πρόγραμμα περιφερειακής συνεργασίας, τα προγράμματα μάλλον περιφερειακής συνεργασίας να εφαρμοστούν με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε επί τη βάση αυτών των τροπολογιών συμβιβαστικέ που να μπορούν να σταθούν και μετά όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ στις τροπολογίες μία προς μία, αλλά ελπίζω πως θα έχω τη στήριξή σας έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό πακέτο. Τώρα, για αυτές τις τροπολογίες υπάρχουν ομαδοποιήσεις, υπάρχουν επικαλύψεις. Είδαμε ήδη πως ορισμένα στοιχεία καλύπτονται από τις τροπολογίες που εγώ ίδια κατέθεσα. Θα αναφέρω τρία χωριστά στοιχεία που ίσως ε, να δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα. Καταρχήν, πολλές τροπολογίες αφορούν την χρηματοδότηση ότι δηλαδή θα πρέπει να γίνεται άμεση χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων. Το έχουμε συζητήσει επανελειμμένως με την, με την Κομισιόν, αλλά θα ήθελα και πάλι να ακούσω την Κομισιόν που θα πρέπει να μας αιτιολογήσει την θέση της και πώς και πού θα μπορούσε να διαβλέψει προβλήματα με βάση αυτές τις άμεσες ε, πληρωμές. Τώρα που έχουν ξεκινήσει δύο διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, συνάδελφοι, θα πρέπει να σταθούμε πολύ στεναρά απέναντι. Εγώ ε, έχω προ... προτείνει το 7% για αυτό το πρόγραμμα προπολογισμού συνοχής. 3,48 ήταν το νούμερο που μας έδωσε η Κομισιόν. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το 7% δεν θα το φτάσουμε, αλλά Εάν επιθυμούμε να διατηρήσουμε τουλάχιστον τρία και κάτι, το Κοινοβούλιο θα πρέπει πραγματικά να παρουσιαστεί πολύ ισχυρό και να απαιτήσει το 7%. Εάν στις διαπραγματεύσεις θέλουμε να στοχε... μάλλον, στοχεύσουμε αρχικά στο 7% θα πετύχουμε το στόχο που αρχικά επέβαλε η Κομισιόν. Αν είμαστε σταθεροί λοιπόν σε αυτό το στάδιο θα τα πάμε καλά. Ξέρουμε ότι τα χρήματα είναι περιορισμένα και ότι ο ελοχεύει ο κίνδυνος ε, να βρεθούμε κάτω από τους στόχους της Κομισιόν όσον αφορά αυτά τα προγράμματα. Επιπλέον, και αυτή είναι η τρίτη μου παρατήρηση, που δίχασε την Επιτροπή μας, 150 χιλιόμετρα είναι το όριο όσον αφορά τα διασυνοριακά εδάφη. Εγώ η ίδια ήμουνα κάπως ε, διστακτική όσον αφορά την ισχύ αυτής της απόστασης ή αυτής της ε, γεωγραφικής περιοχής, γιατί αν μιλάμε για παράδειγμα για νησιά, είναι σημαντικό στην περίπτωση αυτή να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που προβλέπονται από τις, τα διασυνοριακά ε, δάφη, δηλαδή το Strand B, και πρότεινα ανάμεσα στα δήματα Α και Β να μπορούμε να έχουμε ένα περιθώριο ελιγμού της τάξης του 15% πράγμα που θα μας επέτρεπε να μην αποκλείσουμε τις νησιωτικές περιοχές. Όσον αφορά τις, τα υπερπεριφερειακά εδάφη και κτίσεις, πολλές δυνατότητες παρουσιάστηκαν ήδη. Αυτές ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές έχουν ε, ήδη μπορέσει να εκμεταλλευτούν τα κονδύλια ακόμα κι αν ε, υπερεύναν τα 50 χιλιόμετρα. Είμαι πολύ προβληματισμένη όσον αφορά την αύξηση αυτής της απόστασης 100, κατά 100 χιλιόμετρα και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να βρούμε ε, μια συμβαστική λύση και για αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φρανσέσκο Δεντζέλης. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι πολλές από τις 370 τροπολογίες που υποβλήθηκαν είναι τροπολογίες που ακολουθούν τη σωστή πορεία. κυρίως το στόχο μιας ε, πιο φιλόδοξης εδαφικής συνεργασίας, η οποία να ενσωματώνει κυρίως ε, τα στοιχεία της κοινωνικής ισότητας. Πιστεύω λοιπόν ότι ως προς αυτό είναι θετικές οι τροπολογίες της Περβάνς Μπερέζ, που έρχονται από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων διότι είναι τροπολογίες πολύ σημαντικές. που κυμαίνονται από την οικονομική και κοινωνική ένταξη στις μειονεκτούσες περιοχές, στους στόχους 2020 και κυρίως στην διαφάνεια της αγοράς και στην κινητικότητα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρίως επειδή είχε τη διάθεση να αναζητήσει ισορροπημένες λύσεις και να συνθέσει τις διάφορες προτάσεις που υποβλήθηκαν. Γρήγορα θα ήθελα να αναφέρω κάποια θέματα. Το πρώτο το υπογράμμισε και η ίδια η συγχύτρια και αφορά το θέμα των κονδυλίων, του προπολογισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση, την δυσχερή και την κατάσταση κρίσης. Κρίση εξαιρετικά δύσκολη, πολύ περίπλοκη, που βαραίνει, πιέζει τους προϋπολογισμούς. Είναι τυχαίο. Υπάρχει και μια απόφαση των ε, διάσκεψη των Προέδρων που ζητά να μην αμφισβητηθούν και να μην συζητηθούν οι δημοσιονομικές πτυχές ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει γιατί σε κάποιες επιτροπές ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις σχετικά με το συγκεκριμένο σημείο. Πιστεύω λοιπόν ότι αν ο στόχος μας ε, είναι να, 7% είναι να προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε το ποσοστό που όρισε η Κομισιόν, θεωρώ ότι είναι σκόπιμη και θετική αυτή η πρωτοβουλία. Ωστόσο, προσέχοντας πάρα πολύ μέσα στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης να μην αφαιρέσουμε πόρους από άλλους στόχους. Γιατί διαφορετικά δεν θα κάνουμε τίποτα, θα κάνουμε μία τρύπα στο νερό. Και εδώ χρειάζεται λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ τις ισορροπίες. Δεύτερο θέμα. Αυτό που αφορά το κονδύλι για την τεχνική αρρωγή. Εμένα δεν με πείθει ιδιαίτερα το συγκεκριμένο σημείο, για, πολύ απλό, για ένα πολύ απλό λόγο. Και το λέω και από άμεση εμπειρία, τουλάχιστον στη δική μου προηγούμενη θεσμική δραστηριότητα, επειδή χρειάστηκε να διαχειριστώ κονδύλια και κοινωτικούς πόρους, θα σας πω το εξή. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφιερώσουμε υπερβολικούς πόρους στην τεχνική αρρωγή που σημαίνει προσωπικό υποδομή, υποδομή, φορείς κτλ. Εμείς πρέπει κυρίως σε μια φάση κρίσης και δυσκολίας να αφιερώσουμε περισσότερους πόρους στις περιοχές, στις περιφέρειες και στους πολίτες εφόσον θέλουμε να συμβάλλουμε, να ευνοήσουμε προγράμματα, να τα προωθήσουμε, να προωθήσουμε επενδύσεις, πόρους που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη, στην ε, απασχόληση. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα το σκεφτόμουν ίσως μόνο για τις περιπτώσεις όπου αυτές οι παρεμβάσεις τεχνικής αρρωγής θα είναι απόλυτα αιτιολογημένες. Έπειτα, να επεκτείνουμε σε πέντε τους ε, θεματικούς στόχους. Εδώ είμαι θετικός γιατί αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία κυρίως ε, υπέρ της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Και αυτό το συστοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εδώ για την ευελιξία θα πρέπει να κάνουμε κάτι πιο θαραλέο. Να μην ξεκινήσουμε από πάνω αλλά από κάτω. Από τη βάση και από τον βασικό ρόλο που πρέπει να παίξουν οι περιφέρειες. Τέλος. Για μένα είναι πολύ σημαντικό η προτεραιότητα που αναφέρεται στην πολιτιστική και τουριστική κληρονομιά. Γιατί θεωρώ ότι η πολιτιστική και τουριστική κληρονομιά είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Και προς αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να απελευθερώσουμε πόρους. Γιατί είναι τομείς που μπορούν να μας βοηθήσουν να ευνοήσουν την ανάπτυξη, την ανάκαμψη και την απασχόληση. Ευχαριστώ και αυτά είχα να πω. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Φρανσουά Αλφόνση τώρα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια. Γιατί θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε συμβιβασμούς. Συμμερίζομαι τον εισηγητή για το ότι έχει πολύ σημασία η θέση μας να είναι ισχυρή έτσι ώστε η δαφική συνεργασία να αποτελέσει σημαντικό και κατά προτερότητα άξονα της νέας προγραμματικής περίοδου. Το Κοινοβούλιο ήταν πάντα κινητήριος δύναμη και πρέπει να παραμείνει. Σίγουρα κάποιο ποσοστό παραμένει χωρίς πρόσβαση. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα μεγάλο το οποίο μπορούμε να έχουμε ακόμα και αν υπάρχει μεγάλη πίεση για να πιεστούν οι φιλοδοξίες της περιφερειακής πολιτικής. Είναι μια φιλοδοξία δικιά μας για την εδαφική συνεργασία που δεν πρέπει να πιεστεί γιατί είναι κατορισμό η πιο ευρωπαϊκή από όλες τις πολιτικές μας. Είναι η ίδια η ιδέα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που στηρίζουμε με αυτήν. Εκ μέρους της ομάδας μου λοιπόν και πολλών άλλων ευρωβουλευτών από τα νησιά θέλω να πω στον εισηγητή ότι η πρόταση προκειμένου να παρακάμψουμε το πρόβλημα δεν με ικανοποιεί. Έκλεισε το μικρόφωνο του ομιλητή και δεν ανοίγει πάλι. Έλεγα λοιπόν ότι δεν μας ικανοποιεί αυτή η πρόταση του συγκητή γιατί δεν συμβιβάζεται με την ίδια την ιδέα της συνθήκης όσον αφορά τις νήσους. Πρώτα απ' όλα δεν είναι λύση, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο η απόσταση, 150 χιλιόμετρα. Υπάρχει και θέμα επίπεδου. Το νησί μπορεί να έχει πολλές περιφέρειες. Η εδαφική συνεργασία όμως γίνεται από ολόκληρο το νησί, από το ΝΑΤΣ 2 δηλαδή, το επίπεδο αυτό ΝΑΤΣ 2. Έπειτα, όσον αφορά το πνεύμα, ο κανονισμός πρέπει να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Δεν είναι η πραγματικότητα η οποία πρέπει να προσαρμοστεί και να βρει το δρόμο της ώστε να ανταποκρίνεται λίγο πολύ ε, σε έναν κανονισμό. Είναι ευθύνη της Κομισιόν λοιπόν να κάνει μία πρόταση τέτοια που να εφαρμόζεται στις νήσους απευθείας. Είμαστε πολλοί εδώ από τις νήσους που έχουμε κινητοποιηθεί και να ξέρετε ότι θα το ζητήσουμε, το έχουμε ήδη κάνει με ανοιχτή επιστολή προς την Επιτροπή και θα συνεχίσουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερα πράγματα για αυτό το θέμα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο Τζιβλάσεκ, όχι. Όχι. Παρακαλώ, Ρόζα Μαλζή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με τις ε, κυρίες γραμμές του έργου της εισηγήτριας. Θέλω να υπογραμμίσω και εγώ ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Γι' αυτό και υπέβαλα μια τροπολογία η οποία περιλαμβάνει την πρόταση της Επιτροπής των Περιφερειών που λέει να είναι έξι οι προτεραιότητες, να είναι περισσότερες δηλαδή. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας είναι το εξή. Ελπίζω να μπορέσω να πείσω την εισηγήτρια για το ότι το κριτήριο των 150 χιλιόμετρων δεν έχει νόημα. Συμφωνώ με τις εξηγήσει που έδωσε ο συνάδελφος Αλφωσίν, αλλά θέλω να δώσω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η νήσος Ρενιόν ή του Μαυρίκιου, 200 χιλιόμετρα και 700 χιλιόμετρα είναι το επόμενο έδαφος που βρίσκεται κοντά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το κριτήριο δεν έχει νόημα και ότι τελικά εμποδίζει τα παράκτια διαμερίσματα και δάφη να αποφεληθούν από θετικά μέτρα για την εδαφική συνεργασία. Ελπίζω λοιπόν στους συμβιβασμούς να μπορέσουμε τελικά να πείσουμε την εισηγήτρια η οποία προ το παρόν είναι σκεπτική, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο σκεπτικισμός της αυτός θα γίνει πεποίθηση μεθαύριο. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Δεν βλέπω να θέλει κανένα άλλο το λόγο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ο Νίκολας Μάρτιν από τη Γενική Διεύθυνση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα επικεντρωθώ σε κάποια από τα στοιχεία κλειδί που αναφέρονται στις τροπολογίες τις οποίες θίξατε σήμερα. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν περισσότερες τροπολογίες για τον κανονισμό ETC παρά για το CPR. Συνεπώς, η θεματική συγκέντρωση. Για μας Επιτροπή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την εδαφική συνεργασία όπως έχει και για άλλα προγράμματα. Και αυτή είναι η βάση, αν θέλετε, για την πρόταση της Επιτροπής. Όσον αφορά τα κονδύλια και δεν θέλουμε να αλλάξει η φύση τους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, το που θα πάνε δηλαδή τα κονδύλια στο ETC ε και έχει εξίσου μεγάλη σημασία όπως πώς θα δαπανηθούν τα κονδύλια που πάνε αλλού. Όσον ε, αφορά τώρα τις προτεραιότητες για τις επενδύσεις. Φυσικά και βλέπουμε εδώ πέρα πολλές ε, τροπολογίες που θέλουν να αλλάξουν τις ε, προτεραιότητες. Αλλά προσοχή, μην υπάρξει επικάλυψη με τόσα υπάρχουν ε, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ΕΤΠΑ. Η εδαφική συνεργασία, μην ξεχνάτε ότι μόνο από την περιφερειακή ανάπτυξη χρηματοδοτείται. Ίσως πρέπει να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά χρειάζεται αποσαφήνιση το πράγμα. Ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί για το εξή. Θέλετε να συμπεριλεύουμε στο επίπεδο των προτεραιοτήτων ή των αντικειμενικών στόχων ε, κάποια μνήμα για τον τουρισμό ή τον πολιτισμό. Ε, μας μας απασχολεί αυτό όχι γιατί λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Φυσικά και πρέπει να υπάρξουν, αλλά πρόκειται για τομείς και όχι για στόχους αυτούς καθεαυτούς. Άρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν με άλλους τρόπους που έχουν να κάνουν με την οικονομική ανάπτυξη κλπ. Νομίζω δηλαδή ότι δίνουμε στραβό μήνυμα όταν μιλάμε για αυτούς σε σχέση με άλλους, ε, με άλλους τομείς. Τώρα και κάποια πράγματα τα οποία δεν αναφέρθηκαν σήμερα, αλλά που υπάρχουν στις τροπολογίες. Για παράδειγμα, για τους σπόρους. Εμείς ε, εμένουμε στις απόψεις που είχαμε και για την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή να γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χορηγηθούν τα κονδύλια κατευθείαν ένα πρόγραμμα. Κυρίως επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία που να διέπονται από αρκετή συνοχή στα διάφορα επίπεδα. Έπειτα ο σχεδιασμός των διαφόρων τομέων, ναι, μεν επιτρέπει και προβλέπεται στον κανονισμό κάποια ελαστικότητα και γίνονται και συζητήσεις και είναι σημαντικό να γίνονται και να αποτελούν και το σημείο κίνησης για από εδώ και πέρα. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να φροντίσουμε οι διάφοροι τομείς ε, του προγράμματος να είναι πιο αποτελεσματικοί. Τώρα το θέμα των 150 χιλιόμετρων. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη ευαισθησία για αυτό το ζήτημα. Σας υπενθυμίζω όμως ότι η εδαφική συνεργασία σχεδιάστηκε με διάφορα στοιχεία. Έχουμε το διασυνοριακό, έχουμε το διακρατικό. Το διασυνοριακό έχει να κάνει με ένα πραγματικό θέμα. Αν δείτε δηλαδή τα χερσαία σύνορα, εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε διάφορα ζητήματα. Μερικές φορές υπάρχει τεχνητός χωρισμός και ανάλογα κατανέμονται και τα κονδύλια. Χρειάζεται κάποιος εξορθολογισμός, όπως επίσης και στα θαλάσσια σύνορα. Δεν μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για σύνορα με τον ίδιο τρόπο, είτε πρόκειται για απόσταση μεταξύ δύο εδαφών που είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα ή όχι. Γι' αυτό θέλουμε να κρατήσουμε το status quo για τα 150 χιλιόμετρα, αλλά τα σχετικά εδάφη δεν αποκλείονται από την εδαφική συνεργασία, διότι είναι και θέμα διακρατικής συνεργασίας. Το θέμα τώρα του προπολογισμού, το δημοσιονομικό. Μας άρεσε αυτό που ακούσαμε από την εισηγήτρια, άρα νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό διαπραγματευτικό δρόμο για το 7%. Η πρόταση της Επιτροπής ήδη μιλάει για μια αύξηση του 30%. Αλλά πρέπει να δούμε και την αποτελεσματικότητα από εμπειρία πρέπει να δούμε ποια είναι τα επίπεδα χρηματοδότησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας. Πρέπει να μπορεί να υπάρχει απορρόφηση. Η ισορροπία πρέπει να υπάρχει όσον αφορά τους όγκους των χρημάτων που πάνε στην εδαφική συνεργασία και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να απορροφηθούν πραγματικά τα κονδύλια αυτά. Η εισηγήτρια, κυρία Μάνερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις και τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις. Για το θέμα του προϋπολογισμού. Είμαι ικανοποιημένη και θα είμαι πολύ ικανοποιημένη αν επιτύχουμε το 7%. Θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις και θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να επιτευχθεί το ποσοστό αυτό. Πρέπει να δούμε όμως ποιες είναι και οι εμπειρίες. <clears throat> βλέπω ότι έχουν διαγραφεί ορισμένα πράγματα από τις προτάσεις της Κομισιόν. Επειδή είναι δύσκολη τώρα η δημοσιονομική κατάσταση, φοβούμαι ότι θα γίνουν και άλλες περικοπές. Πρέπει να είμαστε, να επαγρυπνούμε στο Κοινοβούλιο για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Τα 3,5% κάτι είναι. Γι' αυτό να επιμείνουμε εμεί το 7% ώστε να μην κατέβουμε περισσότερο. Τώρα για τις τεχνικές ενισχύσεις. Είμαι ανοιχτή για το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων. Μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμβασμό, να τονιστεί ιδιαίτερα η ανάγκη αυτή της τεχνικής στήριξης και βέβαια με ιδιαίτερη έμφαση στα μικρά έργα. Τώρα για τα 150 χιλιόμετρα. Αυτά προκάλεσαν αρκετές συζητήσεις. Εδώ τίνω να συμφωνήσω με την Κομισιόν. Πρόκειται εδώ για θέματα διασυνοριακής συνεργασίας. Και η στόχη είναι σαφής. Η διασυνοριακή συνεργασία βέβαια προ, προϋποθέτει ότι συνεργάζονται περιοχές που είναι κοντά στα σύνορα. Και 300 και 400 χιλιόμετρα να το βάλουμε το όριο, πάλι ορισμένοι δεν θα ικανοποιούνται. Τώρα, για τις υπερπεριφερειακές περιοχές θα πρέπει να έχουμε κάποια ευκαμψία. Και υπάρχουν και τα διεθνικά προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν. Αυτά βέβαια μπορούμε να τα επανεξετάσουμε. Ελπίζω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε σε έναν θετικό συμβασμό. Η Πρόεδρος, κυρία Χίπνερ, ευχαριστώ. Ας κλείσουμε το θέμα αυτό και ας προχωρήσουμε στο 17 του Γιάνν Όλμπριχτ σχετικά με την εξέταση των τροπολογιών. Όλμπριχτ στα αγγλικά. Έχω μερικά στοιχεία στις τροπολογίες που επιθυμώ να σας θέσω υπόψη. Πρώτα, γενική παρατήρηση. <clears throat> Ορισμένοι από τους συνάδελφους μας προτείνουν τροπολογίες για αλλαγή του τίτλου των θεματικών στόχων. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι οι θεματικοί στόχοι περιλαμβάνονται στον γενικό κανονισμό, στον οριζόντιο κανονισμό. Άρα τότε πρέπει να αλλάξουν αυτόν τον κανονισμό και όχι εδώ οι Είμαι υποχρεωμένο να απορρίψω λοιπόν όλες τις σχετικές τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά τώρα τους στόχους του ΦΕΝΤΕΡ. Θα προσθεθούν νέα θέματα τώρα για τις δημογραφικές προκλήσεις και μειονεκτήματα. Και γι' αυτό επαχθέσω ότι είναι σημαντικές οι δημογραφικές στατιστικές. Πάντως εδώ οι βουλευτές προτείνουν προσθήκες άλλων, πολλών άλλων στοιχείων. Εγώ έχω προτείνει μοναχά δημογραφικές προκλήσεις. Προτάσεις που βλέπω εδώ είναι και γεωγραφικές και γεωγραφικά μάλλον και φυσικά μειονεκτήματα. Μα ποια είναι η διαφορά μεταξύ γεωγραφικών και φυσικών μειονεκτημάτων. Και κάτι ακόμα που ίσως οφείλεται βέβαια στην άγριά μου. Αλλά ποιες είναι οι υποπεριφερειακές ανισορροπίες. Ίσως να υπάρχουν εγχειρίδια που να τα λένε αυτά. Διαπεριφερειακά, ενδοπεριφερειακά, καλά. Αλλά υποπεριφερειακές ε, ε, ανισορροπίες, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άλλο βέβαια αν εννοούν intra-regional και όχι infra-regional. Αλλά να με εξηγήσουν τουλάχιστον. Ορισμένοι προτείνουν να μπουν όπως είπα και γεωγραφικά και φυσικά και μη διακρίσεις, δηλαδή αποφυγή διακρίσεων. Ας κατανοήσουν συνάδελφοι ότι αυτά όλα μπαίνουν στο γενικό κανονισμό. Δεν υποχρεώμεθα να περιλαμβάνουμε σε κάθε κανονισμό κάτι το οποίο επικαλύπτει τα πάντα. Αν συμφωνούμε γενικά, <clears throat> δεν είναι αναγκαίο να τα επαναλάβουμε τα πράγματα αυτά στο, σε τούτο εδώ το κανονισμό. Δεν έχω καμιά αντίρρηση να μην υπάρχουν ανισότητες των φύλων, αλλά δεν χρειάζεται. Τώρα, για το, για το πεδίο εφαρμογή. Έγινε μια συζήτηση σήμερα, εκτός αιθούσης, για το ποιος θα πρέπει να λαμβάνει την υποστήριξη. Και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Εδώ πάλι πολλές τροπολογίες για το θέμα αυτό. Και βέβαια για τις παραγωγικές επενδύσεις των μεγάλων επιχειρήσεων κλπ. Αυτό λοιπόν θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο. Άλλο υποστήριξη για προσβάσιμες υποδομές και αυτό αναφέρεται κυρίως σε αναπήρους. Να είναι λοιπόν προσβάσιμες οι υποδομές. Κάτι που υποστηρίζουν πολλοί είναι η συμπερίληψη του τουρισμού. Πάλι εδώ είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, ιδίω για την Κομισιόν. Είναι πολύ έφραστο στοιχείο. Εγώ να εξηγήσω πάντως την αιτιολογία και κυρίως του τουρισμού που είναι ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας σε πολλές χώρες. Όχι μόνο ο αθλητισμός, ο τουρισμός. Υπάρχουν και άλλα που προσθέτουν οι συνάδελφοί μου. στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσθεθούν και οι μικροεπιχειρήσεις και η κοινωνική οικονομία, οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Και αυτές λοιπόν να είναι επιλέξιμες για παραγωγικές επενδύσεις. Να διευκρινίσουμε τι εννοούμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικροεπιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας για να ξέρουμε γιατί πράγματα μιλούμε. Άλλο είναι παραγωγικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη και στις παρεμβάσεις χαμηλού άνθρακα, ε, δουσίου του άνθρακα δηλαδή. Επίσης, υποδομές για τα νερά, για την φροντίδα των παιδιών. Τι πάνε να πει λοιπόν κοινωνική υποδομή ή κοινωνικές υποδομές. <clears throat> Αυτά επίσης είναι ζήτημα που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Πάλι στον τουρισμό μικροεπιχειρήσεις, κοινωνική οικονομία, δηλαδή επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Εγώ προτείνω να διαγράψουμε αυτή τη σημαντική φράση σχετικά με την απαγόρευση επενδύσεων σε βασικές υποδομές στον τομέα των μεταφορών του περιβάλλοντος και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας που υποστηρίζεται πολύ αλλά που νομίζω ότι και εδώ πρέπει να διευκρινιστεί και η Κομισιόν να εξηγήσει τι εννοεί όταν μιλεί για βασικές, μάλλον για υποδομές που καλύπτουν βασικές ανάγκες. Πρόσφατα συζητούσαμε θέματα προμήθειας νερού. Υποδομή παροχής νερού είναι βασική υπηρεσία ή όχι. Για πολλές χώρες μέλη όπως Ισπανία, Πορτογαλία έχω την πληροφορία ότι αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες δυσχέρειες σχετικά με το νερό. Εδώ θα απαγορεύεται λοιπόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό από την στήριξη, γίνεται η πρόταση της κατασκευής πυρηνικών σταθμών. Αυτό που περιλαμβάνεται τώρα είναι η ολοκλήρωση των έργων των πυρηνικών σταθμών. Εδώ η πρόταση είναι να αποκλειστεί η κατασκευή. Νομίζω κανένα δεν πρότεινε κατασκευή, γιατί να αποκλειστεί τότε. Να αποκλειστεί επίσης, να αποκλειστούν μάλλον επίσης μεγάλα έργα οδικών υποδομών και γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Πάμε λοιπόν τώρα από τη βασική υποδομή στον τουρισμό και φτάνουμε στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Είχαμε μέσα τον καπνό. Αν έχουμε τον καπνό, τότε αμέσως έχουμε και άλλη πρόταση, σαν αυτή που σας είπα. Για το άρθρο 4, όπως είπα και πριν, έχει γίνει πρόταση να αλλάξει ο τίτλος και λίγες προτάσεις να αλλάξει το ποσοστό από το 8, το 80 στο 50 και διάφορα τέτοια και να αλλάξει τελείως η θεματική συγκέντρωση. Και επίσης ιδιαίτερες διατάξεις για ε, περιφέρειες που βρίσκονται σε μεταβατική φάση. Τώρα, αλλού υπάρχει η τάση να αναπτυχθούν οι προτεραιότητες για τις επενδύσεις να δοθεί περισσότερο περιεχόμενο δηλαδή στις ε, προτεραιότητες επενδύσεων. Δεν θέλω να τα διαβάσω όλα αυτά που έχω λάβει, αλλά περιλαμβάνεται για παράδειγμα η οικολογική καινοτομία, οι, μεταφορές επιχειρήσεων. Γενικά λοιπόν, άλλο, διαχείριση των νερών, τουρισμός, η οικολογική καινοτομία, καινοτομία στις κοινωνικές υπηρεσίες και άλλα τέτοια. Θα έχουμε και την πρόταση να αλλάξει η θέση των μεταφορών από την 7η να πάει στην 4η και να είναι μονάχα η αστική κινητικότητα εκεί, όχι ολόκληρη, ολόκληρη οι μεταφορές, γιατί αυτό θα καταστεί τελικά υπερβολικά δαπανηρό. Αυτά για τις προτεραιότητες επενδύσεων. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, θα προσπαθήσω να τις περιλάβω στις συμβιβαστικέ τροπολογίες. Επίσης, η αστική διάσταση. Εδώ δεν υπάρχουν πολλές τροπολογίες. Πολλοί ζητούν να καταργηθεί η αστική πλατφόρμα και η λίστα των πόρων. Α, αυτό είναι στο γενικό κανονισμό. Ε, συγγνώμη. Επίσης, πρόσθετη στήριξη για αστικές διασυνδέσεις. Μπαίνουμε όμως τώρα σε μια συζήτηση. Θα έχουμε αυτό το περιβόητο 5% για ολοκληρωμένα ή μάλλον για βιώσιμες αστικές δράσεις. Η πρόταση είναι να περιοριστεί μόνο σε πόλεις μικρών ή μεσαίων διαστάσεων. Αυτή θα είναι η επόμενη μάχη που θα έχουμε να κάνουμε. Εγώ προτιμώ να το αφήσουμε αυτό στη διακριτική ευχέρεια των χωρών μελών. Τι είδου πόλει θέλουν να στηρίξουν. Α μην αποφασιστεί αυτό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση να αυξηθεί από το 5% στο 10% οι βιώσιμες αστικές δράσεις. Νομίζω ότι αυτό το 5% ήταν ένα είδος πιλωτικό σχήμα. Αν όμως διπλασιαστεί θα χαθεί αυτός ο χαρακτήρας και θα είναι δύσκολο οι πόλεις να πάρουν ε, τα χρήματα αυτά από αυτές τις ε, πηγές. Επίσης για άλλα θέματα τώρα, περιαστικά, ε, κοινωνικής ευθύνης κλπ. Εκεί το 0,2 των εθνικών δαπανών. Αυτά όμως πρέπει να τα κρίνει η Επιτροπή να τα προτείνει. Πολλές τροπολογίες αναφέρονται πάλι σε περιφερειακές, περιφερειακά και άλλα μειονεκτήματα, φυσικά μειονεκτήματα κτλ. Θα προσπαθήσω και εδώ να βρω κάποια συμβαστική διατύπωση. Νομίζω ότι γενικά, συνολικά έχω 800 τροπολογίες. Πολλές από αυτές όμως ακολουθούν τις γενικές αυτές κατευθύνσεις που περιέγραψα. Επομένως πιστεύω ότι δεν θα δυσκολευτούμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις διότι νομίζω ότι γενικά συμφωνούμε για το τι θα πρέπει να περιληφθεί στο ΦΕΝΤΕΡ. Πάντως, γενικά έχω την εντύπωση ότι οι ευρωβουλευτές συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει θεματική συγκέντρωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Θεματική συγκέντρωση λοιπόν λέμε ναι. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό, σε ποιο επίπεδο λεπτομέρειας θα πρέπει να μπούμε τι θα πρέπει να υποχρεωτικό και τι όχι, τι θα πρέπει να διαθέτει μια ευκαμψία και τι όχι για τους τελικούς δικαιούχους. Θα συνεργαστώ στενά με τους άλλους συζητητές για να, έχω, να έχουμε μάλλον μια γενική άποψη για τις τροπολογίες και τις συμβαστικές τροπολογίες δηλαδή. Και αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία. Κάτι που είναι σημαντικό και νομίζω ότι δεν υπήρχε στο αρχικό σχέδιο που λάβαμε από την Επιτροπή, από την Κομισιόν, σε σχέση με τον ορίζοντα 2020 δηλαδή. Θα είναι δυνατότητα νομίζω να χρησιμοποιηθούν διαρθρωτικές δαπάνες για την περίπτωση αυτή, αλλά υπάρχει και η τροπολογία που λέμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η σχέση με το CEF Και αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί αυτό το CEF είναι από το Ταμείο Συνοχής. Επομένως, να έχουμε εκτός το ΦΕΝΤΕΡ e e και αυτά. Αυτό είναι αρκετά ευνηδιαστικό. Συνολικά υπάρχουν πολλές τροπολογίες που νομίζω δεν είναι αντιφατικές. Ίσως έχουν διαφορές απόψεων. Τελευταίο σχόλιο θα έχουμε προβλήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυτές είναι από τις πιο μεγάλες διαφορές μεταξύ των πολιτικών ομάδων διότι όλες σχεδόν οι πολιτικές ε, ομάδες λένε ότι θα πρέπει να είναι και για τις μεγάλες επιχειρήσεις εκτός από την ομάδα των πράσινων που λέει όχι μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις τελεία. Εκεί λοιπόν θα έχουμε βέβαια κάποια προβλήματα που πρέπει να διαπραγματευτούμε. Ευχαριστούμε. Γιάννη, πριν ζητήσω από την Κωνστάτσα να πάρει το λόγο, Δελ, αυτό για το infra-intra Ίνφρα σημαίνει μέσα στην περιοχή, ενώ ίνφρα σημαίνει κάτω από το επίπεδο της περιφέρειας. Αλλά θα έπρεπε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας το εξηγήσει παραδοσιακά. Τον όρο ίντρα χρησιμοποιεί, το διά περιφερειακό ας πούμε. Υποθέτω. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι πρόβλημα. Αλλά όντω ας μην το αφήσουμε στους γλωσσομαθείς αυτό, ας το λύσουμε. Δεν ναι, είμαστε πραγματιστές. Κωνσταντ Σακρέλ, λοιπόν, από την Cost Investor. Κυρία Κρέλ, δεν μιλώ ω συντονίστρια, ούτε ω συγγήτρια, αλλά εκπροσωπώντα μόνο την κυρία Βέσφαλ, η οποία κολλείεται σήμερα και η οποία με παρακάλεσε να τα πω για λογαριασμό τη. Πρώτα βεβαίω ευχαριστώ τον Γιάνν Όλμπριχ, τη συγγητή, καθώ και του ε, συναδέλφους. Η ε, κυρία Βέστφαλ εξεπλάγει που για 10 σελίδες καταλήγουν οι συνάδελφοι να γράφουν 800 τροπολογίες. Είναι πάντως μια εμπειρία που γίνεται όλο και πιο συνήθιστα τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες. Η εντύπωση της κυρίας Βέσφαλ είναι πάντως ότι οι βασικοί προσανατολισμοί και των τροπολογιών είναι κοινοί και επομένως θα μπορέσουν να επιτύχουν πλειοψηφία στην ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Για παράδειγμα, για τις τροπολογίες για την ανάπτυξη των ε, υποδομών αλλά και σε πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες θεωρούμε ότι μπορεί να βρεθεί μια συμβαστική διατύπωση που να επιτρέπει την στήριξη επενδύσεων και στις ε, περιφέρειες αυτές. Ο Γιάνν είπε και πριν το πρόβλημα δηλαδή ότι η στήριξη επιχειρήσεων περιορίζεται μοναχά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για πολλές πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, κάπου κάπου καθίσταται αναγκαίο να στηριχθεί και μια κάπως μεγαλύτερη επιχείρηση. Γι' αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται περισσότερο περιθώριο υπέρ των περιφερειών, να έχουν στη διάθεσή τους οι περιφέρειες δηλαδή, για να αποφασίζουν αυτές. Χωρίς να σημαίνει ότι καταρχήν θα είναι πάντα δυνατόν αυτό, έτσι και αλλιώς τα λεφτά δεν φτάνουν για να ε, ε, καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες, αλλά να μπορούν οι περιφέρειες να δίνουν τη δυνατότητα αυτή ενδεχομένως για τη θεματική συγκέντρωση την οποία στηρίζουμε, καταρχήν, πιστεύουμε ωστόσο ότι οι προτάσεις της Κομισιόν είναι κάπως μονόπλευρες και άκαμπτες. Γι' αυτό η δική μας πρόταση κατευθύνεται περισσότερο στην προσθήκη ενός πρόσθετου τέταρτου στόχου και με το ερώτημα αν ενδεχομένως οι περιφέρειες μπορούν οι ίδιες να επιλέξουν τον τέταρτο στόχο που επιθυμούν αναλόγως των αναγκών τους. Εκεί επίσης θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο συμβασμό. Αυτό φαντάζομαι ότι θα μπορέσει να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευση τις επόμενες ημέρες. Ο Γιάνν είπε ήδη ότι πολλοί έχουν ρωτήσει για τα δημογραφικά, για τον τουρισμό, για τον πολιτισμό θεωρούμε ότι ο τουρισμός αλλά και τα πολιτιστικά και η βιομηχανία της δημιουργίας, ας το πω έτσι, είναι παράγοντας ανάπτυξης για πολλές περιφέρειες. Και εδώ είναι σημαντικό λοιπόν να συζητηθεί στα πλαίσια του Περιφερειακού Ταμείου. Επίσης μια υπόδειξη, βεβαίως υποστηρίζουμε στα πλαίσια της μελλοντική πολιτικής συνοχής να προαχθεί και η στρατηγική του 2020. Όμως χωρίς να λησμονούμε τα κλασικά καθήκοντα του Περιφερειακού Ταμείου, όπως τα λέει και το άρθρο 2. Πρέπει αυτό να περιληφθεί και πάλι ρητά, ότι δεν πρέπει να λησμονηθούν οι στόχοι αυτοί. Τώρα, για την στήριξη των αστικών κέντρων είμαστε υπέρ και υποστηρίζουμε μάλιστα τις τροπολογίες για το Φόρουμ Ανάπτυξης των Αστικών Κέντρων, καθώς επίσης να υπάρξει ένας άξονας προτεραιότητας για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, που να συνδέει πολλούς άξονες μεταξύ τους. Κατά τα άλλα, η κυρία Βέστφαλ, την οποία, όπως είπα, πρόσωπο εδώ, δηλώνει την διάθεσή της για συνεργασία για τις επόμενες εβδομάδες, βέβαια με στόχο στις 11 Ιουλίου να υπάρχει ο συμβασμός τον οποίο να μπορούμε να ψηφίσουμε. Ευχαριστούμε. Βλάσακ, ο επόμενος ομιλητής. Δεν έχουμε φιλελεύθερους πράσινους, οπότε εσείς έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Από την αρχή πρέπει να σας πω ότι και εγώ και η ομάδα μου παρατηρούμε στενά τις εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις και τη συζήτηση γενικά που γίνεται για τους κανονισμούς αυτούς. Έχουμε πολλά κοινά σημεία με τον Γιάννα Ολμπρεχτ. Αυτό που με καίει πιο πολύ εμένα είναι η αρχή που λέει ότι όποια ανισορροπία δεν έχει να κάνει με αυτό το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να μείνει απ' έξω. Πρέπει να επικεντρωθούμε στον πυρήνα του ζητήματος και να συμφωνήσουμε για το τι θα συμπεριληφθεί στον κοινό αυτοκανονισμό. Ό,τι δεν εμπίπτει άμεσα σε αυτό, να μην απέξω. Κάποιοι ορισμοί βέβαια πρέπει να διευκρινιστούν παρετέρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, τι είναι παραγωγική επένδυση. Συμφωνήσαμε σε αυτό και στο πρόγευμα εργασίας που είχαμε. Ήμασταν πολύ εκεί. Πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνουν οι διάφοροι όροι. Έπειτα για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον τουρισμό μεταξύ των προτεραιοτήτων. Ναι, και εδώ προτείναμε ένα μεγάλο αριθμό προτεραιοτήτων, αλλά μπορούμε να δεχτούμε ένα συμβιβασμό. Και με το 4 θα συμφωνούσα. Και αν επηρεάζεται, έχει να κάνει με την περιφέρεια δηλαδή μια προτεραιότητα και αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε. Για την αστική ανάπτυξη τώρα. Για μένα όλο και περισσότερη στήριξη χρειάζεται. Ναι, στην πρόταση του 10% θα μπορούσα να συμφωνήσω, αλλά πρέπει να δούμε και πώς ακριβώς θα υπολογίζουμε τις επενδύσεις τι θα συμπεριλαμβάνουμε στις επενδύσεις. Αυτό είναι ένα ελάχιστο ποσοστό. Και θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση και σε κάποιες επιπλέον προτεραιότητες. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τώρα. Αν πρέπει να συμπεριλάβουμε και μεγάλες επιχειρήσεις ή μόνο μικρομεσαίες. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να εξαιρέσουμε καμία επιχείρηση. όπου υπάρχουν προοπτικές για έρευνα και ανάπτυξη. Είναι πράγματα που τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ, τις σχετικές επιχειρήσεις, οπότε υπάρχει συμπληρωματικότητα εδώ με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, πρέπει να διευκρινίσουμε και το θέμα του ΦΠΑ πρέπει να είναι ένα λογικό κόστος για μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης να αντιδράσει σε αυτό για το ΦΠΑ. Ε, Κορνέλη δεν είναι εδώ, Κόβατσεφ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έκθεση του κυρίου Όλμπριχτ και θα προσπαθήσω να περιορίσω τις παρατηρήσεις μου στα κύρια σημεία. Δηλαδή, πώς θα πετύχουμε ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και την ελαστικότητα στην θεματική συγκέντρωση. Αυτό θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες για να καταλήξουμε στους συμβασμούς πριν από την 10η Ιουλίου. Πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα στην Ευρώπη. Μα αρέσει, δεν μα αρέσει, είτε στην Επιτροπή, είτε στο Συμβούλιο ή εδώ. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσουν περισσότερο όσον αφορά τι υποδομέ του για να βρεθούν στο ίδιο επίπεδο με τι πιο ανταγωνιστικέ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την, για την εποχή της καινοτομία αν προηγουμένως δεν βοηθήσουμε να υπάρξει η ανάπτυξη που χρειάζεται. Η πολιτική συνοχής λοιπόν θα πρέπει να έχει έτσι ώστε κάθε φορά που γίνεται μια επένδυση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή χαμηλού άνθρακα αυτό πρέπει να γίνεται παράλληλα και με τη γενικότερη ανάπτυξη. Έπειτα υπάρχει το άρθρο, η τροπολογία στο άρθρο 4 που μιλάει για την ε, χρηματοδότηση σε υποχρεωτικούς θεματικούς στόχους. Ξέρω ότι ακούσαμε για το 40%. Ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό με 35% για παράδειγμα. Αυτό το μέρος, το κομμάτι των υποχρεωτικών επενδύσεων από το Ταμείο το Αναπτυξιακό προς τους θεματικούς ε, στόχους, πρέπει να τα αποκρίνεται, είπαμε, στις ανάγκες των περιφερειών. Άκουσα την πρόταση της κυρίας Κρέλ να δημιουργήσουμε έναν τέταρτο στόχο που θα θέτουν οι ίδιες οι περιφέρειες ανάλογα με τις ανάγκες τους. Εντάξει, οπότε περιμένω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα δουλέψουμε πάνω σε αυτή την ιδέα, θα δουλέψουμε με ελαστικότητα και θα πετύχουμε τους ε, σωστούς συμβασμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βλέπω μπαίνουν διάφορε στην αίθουσα και βγαίνουν. Θέλω να πω στους βοηθούς ότι αν δεν είναι εδώ οι βουλευτές σας, αν μη τι άλλο πάρτε τα έγγραφα μαζί σας, μετά να τους τα δώσετε. Γιατί να ξέρετε ότι οι τροπολογίες δεν θα ξαναμοιραστούν τον Ιούλιο. Μην τις ξεχάσετε. Άννα Μιράντα. Ε, Ευχαριστώ. Σε σχέση με αυτά που λέει ο συγγητής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχουν εδάφη που δεν έχουν μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι γεγονός αυτό. 5.000 απασχολούμενων. Υπάρχουν εδάφη που έχουν 100, 200 ε, απασχολούμενους. Για το θέμα του φίλου τώρα. Δεν είναι επειδή είμαι γυναίκα που το λέω αυτό, αλλά πάντως σε όλα τα έγγραφα των ε, θεσμικών οργάνων πάντα λέμε ότι πρέπει να υπάρχει το streaming αυτό, δηλαδή να υπάρχει παντού σε κάθε έγγραφο, σε κάθε πολιτική η διάσταση του φίλου. Αυτό είναι γνωστό. Για την προσβασιμότητα τώρα στις υποδομές. Για τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Τι είδη προγραμμάτων θέλουμε. Μεγάλα βιώσιμα που να λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον. Δεν είναι απαραίτητα πράσινα προγράμματα. Σε μερικές όμως πόλεις της Ευρώπης υπάρχουν μεγάλα προγράμματα και καταλήξαμε για παράδειγμα να έχουμε την ευρωζηνικότητα και, στο... και στην Ήπεθρο για να ενημερώνεται καλύτερα ο κόσμος, να είναι διαδικτυωμένιος. Για τις κοινωνικές Τώρα υποδομές. Ένα σχολείο, για παράδειγμα, μπορεί να έχει ένα σύστημα ενεργειακής ε, απόδοσης ή ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας, όπως και μια μεγάλη επιχείρηση. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε αυτό τον παραλληλισμό. Τέλος, κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι να διευκρινίσουμε τι είναι οι βασικές υποδομές. Εδώ μέσα για μας τους περισσότερους αυτό είναι σαφές, αλλά όχι για όλους. Νίκολα Μαρτίν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σχολιάσει παρακαλώ όσον αφορά ό,τι θέλετε τέλος πάντων και το EDF και ό,τι άλλο θέλετε. Mm. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξαιρετικά σημαντικό ο κανονισμό, γιατί πρόκειται για το μεγαλύτερο κομμάτι χρηματοδότηση στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή. Και σε αυτόν τον κανονισμό βλέπουμε και τι διάφορε διατάξει για να επιτύχουμε συγκέντρωση και στόχευση της χρήση των πόρων. Η λογική είναι να επιτύχουμε αποτελεσματικότητα όσον αφορά την προσθεθέμενη αξία από κάθε ευρώ που δαπανάτε, που χρησιμοποιείτε από τα χρήματα του EDF για επενδύσεις στα κάτι μελη Και αυτό που βλέπουμε εδώ είναι διάφοροι τρόποι για να το πετύχουμε αυτό. Σημείο κίνηση είναι οι περιορισμοί στο πεδίο εφαρμογής της χρήσης της ιδέας που αναφέρεται εδώ και είναι σημαντικό να το δούμε αυτό και να εξετάσουμε τις προτάσεις ε, τροπολογιών σε αυτό το πλαίσιο. Λόγω αποκλεισμού των επενδύσεων σε μεγάλες εταιρείες στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες είναι γιατί ε, έχουμε δει από αποδείξεις ότι από τα στοιχεία που έχουμε ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να δαπανίσουμε τα χρήματά μας. Καλύτερα είναι να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες και ότι δεν είναι χρήσιμο να τοποθετούμε χρήματα σε μεγάλες επιχειρήσεις. Στι πιο ανεπτυγμένε περιοχές. Αυτός είναι ένας γενικός περιορισμό των επενδύσεων στις μεγάλες επιχειρήσεις όσον αφορά τις παραγωγικέ επενδύσεις, διότι δεν πρόκειται για έναν αποτελεσματικό τρόπο παροχής στήριξης. Αποτελεσματικός τρόπος παροχή στήριξης για μεγάλες εταιρείε είναι μέσω τη παροχή ενό καλού περιβάλλοντο για την επιτυχία του μέσω δηλαδή τη δημιουργία υποδομών καλά εκπαιδευμένου προσωπικού, εργατικού δυναμικού, αλλά όχι δίνοντας απευθείας χρήματα. Δεν είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος στήριξής τους. Ο άλλος περιορισμός πεδίο εφαρμογής ε, που ισχύει για τις πιο αναπτυγμένες ε, περιφέρειες όσον αφορά τις επενδύσεις για υποδομές που σχετίζονται με τις βασικές υπηρεσίες, η λογική εδώ είναι ότι οι περιορισμένοι όγκοι χρηματοδότησης στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές δεν δαπανώνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υποδομών, για την κατασκευή δρόμων, σιδηροδρόμων, ε, αποχετευτικών συστημάτων. Δεν είναι αυτό αυτός ο στόχος. Ο στόχος θα πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες της Ένωσης, δηλαδή καινοτομία, στήριξη των μικρομεσαίων, επενδύσεων που θα προωθήσουν την ανάπτυξη και θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Είναι τμήμα λοιπόν αυτής της δικασίας διαβούλευσης ότι περιορισμός, θα πρέπει μάλλον να δούμε το περιορισμό του πεδίου εφαρμογής Μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης έπειτα έχουμε το επόμενο στρώμα συγκέντρωσης όσον αφορά τις προτεραιότητες επενδύσεων. Αυτό γίνεται εντοπίζοντας λεπτομερείς στόχους για τη χρήση της σηματοδότησης για να διοχετευθούν οι πόροι στους πιο σημαντικούς στόχους μέσα στο πλαίσιο των θεματικών στόχων. Και είναι επίσης ε, για αυτό το λόγο που η Κομισιόν έχει ζητήσει να μην αποδυναμωθούν οι στόχοι, ε, να μην προσθεθούν ένα σωρό άλλα πρόσθετα στοιχεία, γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο απομακρυνόμαστε από την αποδοτικότητα. Τελευταίο στοιχείο συγκέντρωση είναι βεβαίω ε, το σύστημα των ποσοστών που εξασφαλίζει ότι ένα μίνιμουμ ποσοστό των κονδυλίων ε, χρησιμοποιείται για τους ε, θεματικούς στόχους κλειδιά που έχουν εντοπιστεί για την χρήση των κονδυλίων του EIDF. γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα του συστήματος συγκέντρωσης που προτείνουμε. δούμε λοιπόν τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί εδώ, έχουμε διάφορα επίπεδα αποδυνάμωσης. Και αν όλα αυτά τα προσθέσουμε στους διάφορους μηχανισμούς, καταλήγουμε χωρίς να επιτύχουμε αυτό το βασικό, τον κεντρικό στόχο. Χάνουμε δηλαδή τη συγκέντρωση. Για τις πόλεις να πω ότι η Κομισιόν συμμερίζεται απόλυτα την άποψη του εισηγητή ότι ο κατάλογος των πόλεων και ο εντοπισμό των πόλεων σε σχέση με το 5% θα πρέπει να θεθεί στα κράτη-μέλη. Έχουμε ήδη σαφώς πει όσον αφορά την πρόταση της Κομισιόν ότι η Κομισιόν στηρίζει μια προσέγγιση που δεν προβλέπει απαρίθμηση των πόλεων στο πρόγραμμα αλλά το αφήνει να το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη σύμφωνα με μια μέθοδο ή ένα σύνολο αρχών που θα αναφέρονται μέσα στο πρόγραμμα. Πάντως τα κράτη-μέλη θα είναι αυτά που θα πρέπει να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση αυτή. Έρχομαι τέλος σε ένα-δύο πιο συγκεκριμένα ερωτήματα που έγιναν. Το ΦΠΑ δεν καλύπτεται σε αυτόν τον κανονισμό. Είναι ένα θέμα το οποίο καλύπτεται στον κανονισμό περί γενικών διατάξεων, γιατί ακριβώς θέλουμε να έχουμε κοινό κανόνα για το ΦΠΑ για όλους ε, τις ε, δραστηριότητες της Κομισιόν και όσον αφορά την ανάπτυξη της υπέδρου, την αλληλεία. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει αυτό για όλα τα κονδύλια, γιατί είναι λογικό, εξασφαλίζει τη συνοχή και διευκολύνει τη ζωή των δικαιούχων και των διαχειριστών των προγραμμάτων. Γι' αυτό και η Κομισιόν έχει προτείνει ε, κάτι που κατά τη γνώμη της ήταν ισορροπημένο. Επιτρέπει την χρήση του ΦΠΑ μόνο σε περιπτώσεις όπου δεν γίνεται να ανακτηθεί, ε, μάλλον επιτρέπεται να μετρηθεί ως δαπάνη. Γιατί διαφορετικά ε, δεν θα πρέπει να φεύγει η ΦΠΑ από, το κοινοτικό, από τα κοινοτικά κονδύλια και να καταλήγει στις, ε, στα εθνικά θησαυροφυλάκια. Γι' αυτό και προσθέσαμε μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο αποκλεισμό για τις υποδομές. Γιατί στο παρελθόν μη δημόσια όργανα δημιουργούνται ειδικά ώστε να μπορέσουν να παρακάμψουν τον κανόνα ΦΠΑ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να είναι δυνατόν. Για το θέμα του, του διαπεριφερειακού και του ενδοπεριφερειακού. Να πω ότι το η διαπεριφερειακό είναι μια ορολογία που ευρέως χρησιμοποιείται σε περιστάσεις εσωτερικής, εσωτερικών περιφερειών. Το υπόλοιπο είναι υποπεριφερειακό, ένδοπεριφερειακό ε, και χρησιμοποιείται γενικά όσον αφορά το θέμα της πολυπίπεδης διακυβέρνησης. Μιλάμε δηλαδή για υποπεριφερειακά επίπεδα στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, για παράδειγμα, και εννοούμε με αυτό τους Δήμους. Ένδο περιφερειακά, δεν, περιφερειακά δεν νομίζω να έχει χρησιμοποιηθεί ως όρος. Βασικές υποδομές και παραγωγικές επενδύσεις και εδώ είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ε, κάποια βάση και πηγές για όλα αυτά. Το ακούσαμε και στη σημερινή πρωινή συζήτηση όπου έγινε αναφορά στις παραγωγικές επενδύσεις και εκεί υπέδειξα πως και αυτό, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται ε, όσον αφορά μια αρχική επένδυση και την κρατική σχετική ορολογία. Πρόκειται για επενδύσεις, για κεφάλαια που συνδέονται με πρωτογενή παραγωγή και που χρησιμοποιούνται από κάποια εταιρεία. Θα κοιτάξουμε να σας δώσουμε πάντως κάποιο υλικό αναφοράς ε, όσον αφορά τη χρήση αυτής της ορολογίας. Αν κάτι τέτοιο σας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία κατά τις επόμενες μέρες ε, στην προετοιμασία των ε, συμβαστικών τροπολογιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Ιαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε μια μακρά συζήτηση με την Κομισιόν για την θεματική συγκέντρωση. Και νομίζω πως η βασική διαφορά που έχουμε με την Κομισιόν και που προκύπτει από πολλές τροπολογίες που έχουμε συγκεντρώσει είναι ο τρόπος με τον οποίο νοούμε την ευελιξία. Γιατί αυτό που προτείνει το σχέδιο της Κομισιόν είναι να εστιάσουμε στα, σε πολύ συγκεκριμένους ε, τρεις θεματικούς στόχους. Τελεία. Και μετά μπορούμε να συζητήσουμε τα ποσοστά που θέλουμε. 20, 50, 60 δεν έχει σημασία. Και μετά να συζητήσουμε το περιεχόμενο. Το κρύβεται πίσω από τη θεματική συγκέντρωση. Η άλλη προσέγγιση είναι να υποχρεώσουμε τους τελικούς δικαιούχους να συγκεντρωθούν οι ίδιοι και να τους δώσουμε σε αυτούς τη δυνατότητα να αποφασίσουν τι είδου συγκέντρωση είναι η καλύτερη ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής 2020. Αυτή είναι η τελική συμφωνία εταιρική σχέση, ανάπτυξη, ε, ε, μάλλον η πέτηση από την Κομισιόν ότι πρέπει να πετύχει του στόχους πρέπει να συγκεντρωθεί, να συγκεντρώσει τους στόχους, αλλά με ποιον τρόπο δεν το λέει. Το ίδιο έχουμε και με την εδαφική συνεργασία. Δίνουμε τέσσερις θεματικούς στόχους και λέμε ότι πρέπει να επιλέξετε τους τρεις. Αλλά αυτό σημαίνει πως εσείς είστε υπεύθυνοι. Πρέπει να αποφασίσετε για το πώς θα επιτύχετε τους στόχους αυτούς. Σήμερα είναι σαν να λέμε δηλαδή, εμείς ξέρουμε καλύτερα τι είναι καλό για σας. Μιλάμε για 20%, 30%, τα, είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι όντως πιο ξεκάθαρα, αλλά ο κανονισμός δεν είναι το, ο στόχος, δεν είναι ο σκοπός, είναι η αρχή. Και μετά έχουμε τα προγράμματα, τι διαπραγματεύσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση για τις ε, παρεμβάσεις τους, τις παρατηρήσεις τους. Ήταν πολύ θετικές. Στην ουσία έχουμε τις ίδιες απόψεις, ακόμα και αν ε, δεν συμμεριζόμαστε απόλυτα όλες τις λεπτομέρειες. Εάν πάντως, ε, όπως είπατε, σε κάποια περιοχή δεν υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, υπάρχουν μικρές. Καλύτερο είναι να πούμε μικρές ή μεγάλες. Ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει. Γιατί δεν βρισκόμαστε σε ένα νησί. Εντάξει, δεν μιλάμε για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει στο Συμβούλιο. Δεν είμαστε απομονωμένοι. Ξέρουμε πώς αλλάζουν τη θέση τους. Γίνονται όλο και πιο ευέλικτοι. Πολλέ από τι τροπολογίε είναι αντικατοπτρισμοί των θέσεων του Συμβουλίου, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε τι συμβαίνει εκεί. Το Συμβούλιο είναι έτοιμο να ανοιχτεί περισσότερο και να μην πει όχι στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά να πει εν γέννη είναι καλύτερο να δίνουμε στις μικρομεσές, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να επιφεληθούν και οι μεγάλες εταιρείες. Και νομίζω θα πρέπει επίση να διευκρινίσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για τουρισμό, πολιτισμό, αθλητισμό. Αυτό δεν θα πρέπει να μπουν βέβαια στον κανονισμό, θα πρέπει να τα συζητήσουμε αργότερα. Πάντως εν γέννη νομίζω ότι συμφωνούμε και ότι θα βρούμε τρόπο να παρουσιάσουμε τη θέση τη επιτροπή μα και Γνωρίζοντας το επόμενο διδικοστικό βήμα, πιστεύω θα βρεθεί τρόπο για να βρούμε συμβιβασμό και με την Κομισιόν ώστε να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά όλα αυτά. Τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι όλοι μας, τα μέλη του Κοινοβουλίου, ξέρουμε πάνω κάτω τι συμβαίνει και προσπαθούμε να τα καταστήσουμε όλα αυτά σαφή για τους ε, δικαιούχο. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση, να φτιάξουμε ένα κείμενο νομικό το οποίο να είναι σαφέ για όλους, όχι για τις κυβερνήσεις, αλλά για όλους. Να είναι όσο γίνεται πιο απλό. Ας το πούμε απλοποίηση. Αλλά απλοποίηση σημαίνει, συνήθως καταλήγει σε περισσότερη περιπλοκότητα. Ας το καταστήσουμε σαφέστερο λοιπόν και πιο ευνόητο. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Πριν περάσω στην επόμενο σημείο που είναι το Ταμείο Συνοχής και ο Βίκτρο Βοστινάρο, θα ήθελα να σα ενημερώσω για τις αποφάσεις που ελήφθησαν εχθές από τους συντονιστές. Ε, δώσαμε νομοθετικές και μη νομοθετικά έγγραφα στις πολιτικές ομάδες, τα αναθέσαμε. Η Άλντε αποφάσισε να πάρει την ειδική έκθεση για τα διευθυντικά ταμεία και τις ελλείψεις τους. Μια άλλη έκθεση για την ΕΛΤΑ είναι μια ειδική έκθεση για τη χρήση των διαθετικών ταμείων και ταμείων συνοχής για την βελτίωση υποδομών στα λιμάνια. Επίσης ε, διατάξεις ε, για τα γεωργικά προϊόντα και οι σοσιαλδημοκράτες, βελτίωση της πρόσβασης στην οικονομία, ΕΛΚ, ενεργειακό οδικός χάρτης 2050 και επίσης ξεκινήσαμε συζήτηση για τις εξωτερικές μελέτες ε, που έχουμε τη δυνατότητα να αναθέσουμε, διότι υπάρχει σχετική χρηματοδότηση και αναμένω πριν από το καλοκαίρι τις αποφάσεις της πολιτικής ομάδας για το τι είδος ε, ε, εξωτερικές μελέτες θα χρειαστούμε. Τελευταίο θέμα θα το συζητήσουμε με τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης που θα κάνουμε στο δεύτερο ήμιση του έτους. Συμφωνήσαμε ότι η αντιπροσωπεία στην Ισπανία, στα Ισπανογαλλικά σύνορα θα γίνει στην εβδομάδα 24, στην Κύπρο την εβδομάδα 39 και μέχρι το τέλος του μήνα όλες οι πολιτικές ομάδες είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν για τον αριθμό των μελών τους που θα πάνε στην Κύπρο, Ισπανία και Γαλλία και ελπίζουμε πως θα έχουμε χρόνο να οργανώσουμε ακόμα μια αναποστολή στην Ιρλανδία. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς οι συνάδελφοι θα αποφασίσουν να πάνε στην Κύπρο και στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Βίκτορο Μπουστινάρο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μόνο 103 τροπολογίες έχουν υποβληθεί για τον κανονισμό αυτό. Αν το συγκρίνουμε με την κατάσταση σε άλλες ε, εκθέσεις, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Βέβαια πήρε χρόνο η μετάφραση και έτσι άργησαν οι μεταφράσεις να είναι διαθέσιμες. Τώρα όμως τις έχετε. Έχω να κάνω κάποια γενικά σχόλια για την εκθεσία μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ επειδή η γραμμή που ακολουθώ στηρίζεται από ό,τι φαίνεται από τους συναδέλφους. Πολλές από τις τροπολογίες μου μάλιστα ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις δικές σας προτάσεις. Είναι πολύ κοντά. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι θα πετύχουμε μια καλή λύση και καλούς συμβιβασμούς πάνω στους οποίους θα βασιστούμε για τη συνέχεια που θα ικανοποιούν όλες τις πλευρές. Πολλές τώρα τροπολογίες είναι προκειμένου το Ταμείο Συνοχής να γίνει πιο πράσινο. Όντως αυτό ήθελα κι εγώ, να πρασινίσει λίγο. Αλλά χρειάζονται πολλά βήματα βέβαια και για τις υποδομές, για τις μεταφορές προκειμένου και αυτές να μπορούν να επιλεγούν για χρηματοδότηση από το Ταμείο αυτό. Η ιδέα πάντως του Ταμείου Συνοχής να χρηματοδοτήσει και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε. Και οι τροπολογίες εκείνες οι οποίε θέλουν να διευρύνουν ε, το εύρο εφαρμογή. πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι αν το κάνουμε αυτό πρέπει τότε να τροποποιήσουμε το άρθρο 9 του τρέχοντος κανονισμού. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες για την ε, μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Ξέρετε ότι είμαι κατά μια τέτοια αρχής. Οπότε, η δικιά μου υπεποίθηση είναι να κρατήσουμε τους τρέχοντες κανόνες της Λισαβόνας στο Ταμείο Συνοχής. Αν το κάνουμε αυτό, θα το δεχτούν όλοι νέες μακροοικονομικές αιρεσιμότητες καταλαβαίνετε θα αποτελούν ε, μια τιμωρία για τις περιφέρειες και τους δήμους πρώτον και δεύτερον θα οδηγήσουν σε διακριτική εφαρμογή των όρων αυτών σε σύγκριση με άλλα κονδύλια συνοχής. Τώρα, όσον αφορά τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Είναι πράγματα τα οποία έχουν συζητηθεί πάρα πολύ, αλλά δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Η δικιά μου άποψη είναι σαφής. Την ξέρετε. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για μένα. Εδώ πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε για να μπορούμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά τα μέτρα, δεύτερον να αποφύγουμε νέες εντάσεις, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν εντάσεις και διαφωνίες μέσα στο Συμβούλιο. Δεν είναι αλήθεια ότι το Συμβούλιο Μεταφορών έχει καταλήξει σε συμφωνία για τη χρηματοδοτική διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Στο Βουκουρέστι συζητήσαμε και με τον κύριο Παρόσο και ξέρουμε ότι 14 χώρες μέλη έχουν ε, δηλώσει ή ότι είναι κατά ή ότι θέλουν να καλύπτονται οι ανησυχίες τους μόνο τότε. Οπότε κάνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει ελαστικότητα και να κατανοήσει ότι εάν έχουμε πόλεμο στο Συμβούλιο, τότε τίθεται σε κίνδυνο το όλο σχέδιο. Γι' αυτό και προτείνω μια συμβαστική τροπολογία η οποία καθισχάζει και τις δύο ανησυχίε και τα εθνικά κονδύλια και βελτιώνει τις ε, ικανότητες και μετά από τρία χρόνια τότε τα χρήματα μπορούν τελικά να μεταφερθούν σε μια κεντρική διαχειριστική αρχή των Βρυξελών. Μπορεί να μην είναι η ιδανική λύση, συμφωνώ, αλλά πρέπει να καταλήξουμε σε συμβασμό. Και αυτό είναι το μήνυμα που έχω να στείλω και στην Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο και στη Γενική Διεύθυνση μου, διότι αλλιώς, όπως καταλαβαίνετε, το πρόγραμμα δεν θα προχωρήσει. Ο χρόνος περνάει. Το ρολόι και οι δείχτες προχωράνε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι μέχρι τον Ιούλιο. Ας καταλάβουμε λοιπόν για ποιο λόγο πρέπει να καταλήξουμε σε συμβασμό. Εγώ είμαι έτοιμος να δουλέψω προς αυτή την κατεύθυνση του συμβασμού. Ξέρετε ότι εγώ έχω καταθέσει την τροπολογία μου, μια παρόμοια όπως του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής, όπως και για τη γενική εφαρμογή. Έρχομαι τώρα στα κύρια σημεία. Ενέργεια, εξοικονόμηση ενέργειας από τα νοικοκυριά. Δεν υπάρχει αντίρρηση από ό,τι έχω δει. Και χαίρομαι που από ό,τι ακούω και το Συμβούλιο έχει καταλήξει σε συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις όσον αφορά την ε, επιλεξιμότητα για αυτή την εξοικονόμηση ενέργειας. Έπειτα, άλλα προγράμματα ψήξης για παράδειγμα. Από ό,τι φαίνεται πάλι υπάρχει μια κάποια συμφωνία. Αλλά όσοι έχουν καταθέσει τροπολογίες να ξέρουν ότι θα με έχουν κοντά τους για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συνεκτική λύση που να τους καλύπτει και αυτούς. Για τους κοινού δείκτες, άλλες τροπολογίες. Εδώ το έχω εξηγήσει λίγο πολύ. Εμείς στη συνοχή αποφασίσαμε ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει εφαρμοστικές πράξεις για τους καινούς δείκτες. Το ίδιο ισχύει και για το Αναπτυξιακό Ταμείο και για το ECD. Και θα έλεγα στους πράσινους να λάβουν υπόψη τους μια τέτοια λύση, η οποία είναι αποτελεσματική, βιώσιμη και μας βοηθάει να αποφύγουμε άλλες διαφωνίες προσθέτοντας τροπολογίες σε θέματα τα οποία είναι καθαρά τεχνικά ή έχουν να κάνουν καθαρά με στοιχεία. Αυτά στα αφήσουμε στην Κομισιόν. Τι άλλες προτάσεις υπάρχουν εδώ στην εκθεσή μου. Α, τις υπόλοιπες τις στηρίζουν οι συνάδελφοι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το δείχνετε αυτό και με τις τροπολογίες σας. Τέλος, θέλω να πω στους και εισηγητές, αλλά και σε όλους τους συναδέρφους ότι είμαι πεπισμένος πως στο τέλος, εφόσον έχουμε υπόψη μας το πνεύμα που ήταν ανοιχτή συνεργασία μεταξύ μας, ο κανονισμός για το Ταμείο Συνοχής θα υιοθετηθεί με μεγάλη πλειοψηφία, κάτι το οποίο θα είναι ένα πολύ καλό μήνυμα όταν θα λάβουμε και την εντολή διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ και πάλι και είμαι στη διάθεσή σας προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για συμβιβασμούς και έτσι να μπορέσουμε τον Ιούλιο να ξέρουμε πώς είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ, Βίκτορ. Η κυρία Ματσόνη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Δίχως ε, άλλο, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουστινάρο και να του πω ότι συμφωνώ μαζί του όταν ε, λέει ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε την έκθεση αυτή. Και αυτό χρησιμοποιώντας τις ιδέες όλων. Δεν είναι ιδιαίτερα επίμαχο νομίζω το θέμα. Γιατί εγώ προσπάθησα και κατάφερα να υποβάλω ελάχιστες τροπολογίες. Έξι συνολικά. Και γιατί, γιατί θεωρώ έτσι μπορώ να εκφράσω αυτό που είχα πει και άλλη φορά στην Επιτροπή μας, αλλά και στις διάφορες συναντήσεις που είχα τους τελευταίους μήνες με τον εισηγητή. Η μόνη καινοτομία της πρότασης της Κομισιόν είναι το περίφημο αυτό ταμείο, CF. Αλλά ο γενικός κανονισμός του δεν με πείθει. Μιλάει για μια διαδικασία η οποία επιτρέπει την χορήγηση των κοδηλίων αλλά Το θέμα είναι κατά πόσο το δικαίωμα αυτό είναι εθνικό. Εννοείται ότι πρέπει να ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την σωστή χορήγηση των κονδυλίων αυτών. Πιστεύω ότι συμφωνεί και ο κύριος Μποστινάρο με αυτό. Όσο για τους άλλους, για τις άλλες τροπολογίες, ο στόχος είναι να επιμένουμε σε κάποια σημεία. ιδιαίτερα για στη μεταβατική περίοδο προς μια οικονομία χωρίς άνθρακα, χωρίς διοξίδιο του άνθρακα μάλλον, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών. Προσπάθησα να το δω εγκάρσια αυτό, ακριβώς για να λαμβάνετε υπόψη σε όλες μας τις δράσεις. Και έπειτα τελευταία παρατήρηση. Κάποια τροπολογία μου έχει ως στόχο μία διευκρίνηση. Ότι οι πόροι του Ταμείου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε πρωτοβουλία η οποία συνδέεται με το διευρωπαϊκό δίκτυο. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει αντιστάθμισμα για την χρήση του Ταμείου Συνοχής μέσα στο γενικό πακέτο των διευρωπαϊκών δικτύων. Ο κύριος Μποστινάρο έχει και αυτός υποβάλει τροπολογίες. Ξέρω ότι συνολικά είναι 321 οι τροπολογίες. Σίγουρα πολλά στοιχεία θα βρούμε στις τροπολογίες αυτές για παράδειγμα για τις αρμοδιότητες του Ταμείου Συνοχής. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα. Χρειαζόμαστε σαφήνεια. Χρειάζεται μεγάλη ελαστικότητα πάντως για να δουλέψουμε. Όσον αφορά πάντως τις επενδύσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους των άλλων διαρθρωτικών ταμείων. Όσες χώρες χρησιμοποιούν το Ταμείο Συνοχής πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν και τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία. Έχω δύο λόγια ακόμα και για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, στις κατοικίες. Εδώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χρυσόγελος. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή. Ε, σίγουρα είχαμε μια καλή συνεργασία και κινείται προς σωστή κατεύθυνση, όπως είχαμε πει και στην αρχή η εισήγηση ε, του, κυρίου, ε, του, του εισηγητή. Σίγουρα φαίνεται ότι υπάρχει μια ευρύτατη συμφωνία και σύμπτωση απόψεων στο θέμα της ε, προώθηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον τομέα της κατοικίας. Ε, και συμφωνούμε όλοι ότι μια τέτοια κατεύθυνση είναι και αποτελεσματική από άψη ε, κόστους αποτελέσματος και συμβάλλει στη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και βοηθάει και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και δημιουργεί επαγγέλματα. Και αυτό πρέπει να είναι πραγματικά ένα εργαλείο της πολιτικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνούμε και υπάρχει νομίζω ευρύτη συμφωνία ότι θα πρέπει να περιληφθεί στο, στο κοινωνικό ταμείο η χρηματοδότηση για τις περιοχές φύση Natura 2000 με προτεραιότητες βέβαια επενδυτικές ε, στα θέματα της αποκατάστασης της βιοπικιλότητας ε, και γενικά της ανάκαμψης ε, της, ε, της, του βιολογικού πλούτου που έχει η Ευρώπη. Ε, σε ένα σημείο στο οποίο υπάρχει διαφωνία είναι σε σχέση με τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στο ETS. Ε, είναι πολύ γενική διατύπωση παρόλο ότι ο εισηγητής έκανε προσπάθεια να βάλει μια, αν θέλετε, μια συμβαστική διατύπωση για πιλωτικά προγράμματα είναι ακόμα αρκετά γενική γιατί θα μπορούσε να αυτό να αφορά και μεγάλες επενδύσεις. Επομένως ε, θα πρέπει να το προχωρήσει ακόμα περισσότερο αν θέλετε στο να είναι συγκεκριμένα πιλωτικά προγράμματα για πολύ μικρές επιχειρήσεις ίσως αλλά μην ανοίξουμε τον τομέα αυτό και ονομαστούν πιλωτικά προγράμματα και εφαρμογές οι οποίες δεν θα είναι πραγματικά πιλωτικές. Ε, στα θέματα της ε, αύξησης της ικανότητας του προσωπικού ε, των ικανοτήτων δηλαδή ε, στο θέμα του σχεδιασμού της παρακολούθησης εφαρμογής ε, των προγραμμάτων θα πρέπει να γίνει σαφές ότι αυτό πρέπει να εστιαστεί στα θέματα του προσωπικού που είναι στις περιφερειακές και τοπικές αρχές και στα θέματα της ε, κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για να, να πετύχουμε πραγματικά στα θέματα της κοινωνικής συνοχής και θα έλεγα γενικότερα στα θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης. Πρέπει να το τονίζουμε και να το ε, κάνουμε ακόμα ίσως πιο συγκεκριμένο. Στα θέματα της, ε, των προτεραιτήτων για τις μεταφορές, ε, έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στο θέμα της πρόθεσης αυτό που ονομάζουμε βιώσιμες μεταφορές είναι σίγουρα βιώσιμες μεταφορές και συστήματα που συνδυάζουν διαφορετικά μεταφορικά ε, συστήματα ε, και να συμπεριλάβουν σε αυτό και τα θέματα του περπατήματος και της, ε, της ποδηλασίας και της από κοινού χρήσης αυτοκινήτων, το, το car sharing και το, το car pooling και φυσικά γύρω από ένα κορμό δημόσιων συγκοινωνιών έτσι ώστε πράγματι να προωθεί αυτό που είναι και η πολιτική μας εδώ, η βιώσιμη αστική κινητικότητα και γενικά η βιώσιμη μετακίνηση. Ε, νομίζουμε όμως ότι εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πάλι ότι υπάρχει και ένα σύστημα μεταφορών που χρησιμοποιεί τους υδάτινους δρόμους, είτε αυτή είναι ποτάμια, είτε είναι και ε, θαλάσσιοι δρόμοι. Άρα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, παρόλο ότι στο μυαλό των περισσότερων όταν μιλάμε για κινητικότητα, σκεφτόμαστε ε, τις πόλεις και τα συστήματα μέσα στις πόλεις ή ε, το σιδηρόδρομο αυτοκινητοδρόμους κλπ. Αλλά είναι όμως και υδάτινοι δρόμοι και θα πρέπει να τους περιλαμβάνουμε πάντα στα συστήματα μεταφορών. Ε, στα θέματα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι το πιο πετυχημένο εργαλείο είναι προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα. Δηλαδή και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά κυρίως και στην προσαρμογή της στην... στα νέα δεδομένα, θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην ε, προσέγγιση του οικοστήματος. Υπάρχουν πολλά έργα που μπορούν να γίνουν, πολλέ παρεμβάσει. Προτεραιότητα πρέπει όμω να είναι σε αυτά που αξιοποιούν την προσέγγιση του οικοστήματος. Στην πρόληψη του κινδύνου, την αποφυγή του κινδύνου και στη διαχείριση των κινδύνων. Ε, και αυτό είναι και ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει επίση και στην απασχόληση και στην αποκατάσταση βιοπικιλότητας. Δηλαδή έχουμε συνδυασμένους, συνδυασμένες πολιτικές. Δεν έχουμε δηλαδή πολιτικές που αντιβαίνουν και συγκρούονται με άλλους Στόχου από άλλε πολιτικέ, αλλά εδώ μπορούμε να έχουμε μια συνεκτική πολιτική. Και νομίζω ότι αυτό είναι και θα πρέπει να είναι και το ζητούμενο συνολικά σε μια πολιτική συνοχή, ότι όταν χρηματοδοτούμε με δημόσιου πόρου διάφορα έργα, πρέπει να υπάρχει συνοχή στα αποτελέσματα τα οποία επιδιώκουμε. Ε, έτσι κι αλλιώ δεν είναι και απεριόριστα τα δημόσια χρήματα, άρα θα πρέπει να έχουμε στοχευμένε πολιτικέ. Και τέλο, για δύο θέματα, στα οποία νομίζω ότι και η Επιτροπή Περιβάλλοντο τα υιοθέτησε σε μια έκθεση στην οποία ήμουνα ε, σε τροπολογίες που είχα καταθέσει μαζί με άλλους πράσινους συναδέλφους ε, είναι το θέμα των προτεραιοτήτων στου τομεί της διαχείρισης των απορριμμάτων και στους τομείς διαχείριση του νερού. Από τη στιγμή που έχουμε μια πολιτική και για τα νερά και για τα απορρίμματα που έχει μια ιεράρχηση στόχων, η προτεραιότητα τη χρηματοδοτήση αντιστοίχω πρέπει να εξυπηρετεί αυτού του ιεραρχημένου στόχου. Δηλαδή, και βλέπω ότι νομίζω ότι θα υπάρχει ευρύτατη υποστήριξη και στην Επιτροπή τη δικιά μα, ότι αφού η ιεράρχηση στόχων για τη διαχείριση των απορριμμάτων προβλέπει την πρόληψη, την αποφυγή απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση κλπ και τα εργαλεία τα χρηματοδοτικά πρέπει να ενισχύσουν τέτοιε δράσει. Γιατί βλέπουμε πολύ συχνά, ενώ η πολιτική μα είναι σε αυτή την κατεύθυνση, να χρηματοδοτούνται κυρίω είτε χώροι ταφή απορριμμάτων είτε εγκαταστάσει καύση. Επομένω, τώρα έχουμε ένα ισχυρό οικονομικό εργαλείο το οποίο πρέπει να συνδέσει την πολιτική με την υλοποίηση των προγραμμάτων. Αντίστοιχα στα θέματα του νερού, πρέπει η προτεραιότητά μα να είναι η ενίσχυση τη μείωση τη κατανάλωση και τη πατάλη νερού και κυρίω η αποτροπή διαρροών στα δίκτυα διανομής του νερού, ιδιαίτερα μέσα στις πόλεις. Έχουμε, ενώ γίνονται έργα για την ε, προμήθεια νερού, έχουμε την ίδια στιγμή διαρροές στα δίκτυα του νερού μέσα στις πόλεις που φτάνουν το 30 40%. Άρα λοιπόν είναι λογικό και αποτελεσματικό από κάθε άποψη και οικονομική και περιβαλλοντική να επενδύσουμε πόρους στη μείωση των διαρών μέσα στα δίκτυα και φυσικά στη μείωση της πατάλης νερού μέσα σε όλο τον κύκλο της χρήσης του νερού, είτε αυτό είναι κατοικίε, είτε είναι επαγγελματικές δραστηριότητες κλπ. Και βέβαια η επαναχρησιμοποίηση και η αξιοποίηση των γκρίζων νερών, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και η συλλογή του βρόχινου νερού, κάτι το οποίο έχουμε μεγάλη εμπειρία σε περιοχές της Μεσογείου, αφού είναι εκεί πέρα ένα πόρο πραγματικά πολύ σημαντικό, το οποίο ξέραμε να χρησιμοποιούμε παλιότερα ω κοινωνίε, πρέπει να ενισχύσουμε αυτέ τι δράσει έτσι ώστε το βρόχινο νερό, το νερό τη βροχή, να μπορεί να αξιοποιηθεί ε, και με την υποστήριξη των, ε, χρηματοδοτήσεων, των δημόσιων χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Συνοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. αν επιθυμεί να συμμετάσχει στη συζήτηση. Θα προχωρούμε πολύ γρήγορα σε 10 λεπτά. Ο πρόσωπό θα πρέπει να είναι εδώ. Ο Γιάννη πάλι, Όλμπριχτ. Συγχαίρω βέβαια τον εισηγητή για τις προσπάθειες του, αν με επιτρέπει να πω ότι δεν πρέπει να λησμονήσουμε το πραγματικό χαρακτήρα του Ταμείου Συνοχής. Το Ταμείο Συνοχής που δημιουργήθηκε στην εποχή της συνθήκης του Μάστριχτ είχε ένα ειδικό στόχο. Αυτός ο ειδικό στόχος ήταν να μειώσει τα βάρη των χωρών μελών για να τους επιτρέψει να προετοιμαστούν για το Σύμφωνο Σταθερότητας. Η πρώτη πρόθεση λοιπόν ήταν να συγκεντρωθεί το Ταμείο Συνοχής στο εθνικό επίπεδο και στο περιφερειακό. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο του ε, Ταμείου Συνοχής που είναι σημαντικό. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι μεγάλες επενδύσεις στο περιβάλλον, μεταφορές και τώρα έχουμε την ευκαιρία να, να δώσουμε χρήματα και για την αποδοτική χρήση της ενέργειας, για μικρά κτίρια. Ο, όμως, ο χαρακτήρας του Ταμείου είναι οι μεγάλες επενδύσεις. Και γι' αυτό, όπως είπα πριν, το Ταμείο αυτό αναλαμβάνει και τις μακροοικονομικές κυρώσεις. Παράδειγμα της Ουγγαρίας, πριν από λίγο καιρό. Άρα, να επιμείνουμε στον χαρακτήρα του Ταμείου Συνοχής που αφορά τις χώρες συνοχής, να υπερασπιστούμε τον χαρακτήρα του Ταμείου Συνοχής, να μην νερωθεί, να μην δηλαδή αποδυναμωθεί ο χαρακτήρας αυτός. Γι' αυτό να προετοιμαστούμε για να αποδείξουμε ότι τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται μετά από αναλύσεις στο εθνικό επίπεδο σχετικά με την κατανομή των πιστώσεων και όχι σε επίπεδο ΝΑΤΣ 2. Τα υπενθυμίζω αυτά γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικά. Και δεύτερο, να μην επιτρέψουμε να αποδυναμωθεί το Ταμείο. Δεν είμαστε βέβαια πολύ αριθμοί τώρα εδώ, αλλά το αγμένο μας θέμα εδώ είναι η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, Επιτρέψτε μου να ρωτήσω ίσως μια ρητορική ερώτηση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο Κοινοβούλιο δεν συζητούμε τα νούμερα. Συζητούμε το πλαίσιο. Εκτός του ΣΥΕΦ Είδατε να συζητούμε, ό,τι συζητούμε μάλλον τις αλλαγές του ΑΕΠ, συζητούμε άλλα πράγματα του Ταμείου Συνοχής. Αν λοιπόν δεν έχουμε 300 εκατομμύρια από την πολιτική συνοχής, αλλά 250 θα εξακολουθήσουν να είναι τα, τάξη των 10 δισεκατομμυρίων ή θα είναι 5 ή 4. Υποσχεθήκαμε στους εαυτού μας να μην χρησιμοποιούμε νούμερα εκτός από το CF που φαίνεται να είναι σαν κάτι το καθαγιασμένο που δεν επιτρέπεται να το αγγίξουμε. Πρώτο σχόλιο. Δεύτερο ερώτημα μάλλον. Πάλι προς την Κομισιόν. Εδώ βέβαια λόγω άγνοιας. Αν το CF θα είναι στο 1α του προπολογισμού 40 εκατομμύρια. Αν αυτά ληφθούν από το Ταμείο Συνοχή, θα πάει στο 1Β. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα από το 1Β στο 1Α. Εδώ βέβαια ομολογώ ότι δεν γνωρίζω. Η διευκόλυνση ε, συνδέοντα την Ευρώπη, που θα είναι οργανισμό τη Βρυξέλλη, θα πάρει χρήμα από το 1α. Μπορεί να χρησιμοποιήσει χρήματα από το 1β. Αυτό είναι συγκεκριμένη ερώτηση για την έκθεση αυτή, διότι χρησιμοποιούμε χρήματα από το Ταμείο Συνοχής. Αν ληφθούν τα χρήματα αυτά, εξακολουθεί να είναι Ταμείο Συνοχής ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα φύγουν, θα εξαφανιστούν τα, τα, τα κονδύλια αυτά από το Ταμείο Συνοχής. Είναι σημαντικό για τον κανονισμό αυτό. Και πρέπει να διευκρινιστεί το δυνατόν συντομότερο, διότι αν όχι, τότε θα έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για χρήματα συνοχής και από την άλλη μεριά δεν θα είναι. Να μην λησμονούμε λοιπόν ότι το Ταμείο Συνοχή κατευθύνεται στι χώρε συνοχή και πρέπει βέβαια να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τι διατάξει τη συνθήκη. Ευχαριστώ. Βλάθακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο και πάλι. Σύμφωνο απόλυτα ότι το Ταμείο Συνοχής είναι ένα μεγά, για μεγάλα προγράμματα υποδομών και για το περιβάλλον και δεν πρέπει αυτό να το αποδυναμώσουμε, δεν πρέπει να οπισθοχωρήσουμε. Επίσης ε, θα μου άρεσε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ταμείο για να μπορούμε να καλύψουμε ας πούμε τις διαρροές ε, στο δίκτυο ίδρυυσης, αλλά δεν ξέρω πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό δεν γίνεται. Ε, ε επίσης, ε, καλό θα ήταν να μπορέσουμε να μεταφέρουμε 10 δις, ε, όχι όμως από το Ταμείο Συνοχής για το ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, το ΣΕΦ. Η Κομισιόν, ο Νικόλας Μάρτιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, τα όσα έχουμε να πούμε για το Ταμείο Συνοχής τα έχουμε ήδη ξαναπεί. Ε, όσον αφορά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής, θα πούμε ότι το Ταμείο Συνοχής έχει συγκεκριμένο σκοπό, συγκεκριμένη βάση στη συνθήκη. Δεν ε, προορίζεται για όλα τα κρατημέλη αντίθετα από το ΕΤΠΑ. Ε, είναι για τις χώρες όπου το ΑΕΠ είναι κάτω από το 18% του μέσου όρου ε, το 80% του μέσου όρου και χρησιμοποιείται για πολύ συγκεκριμένους στόχους και η χρήση του δεν θα πρέπει να αλλάχτεί, γιατί να αλλάξει με τρόπο όπως φαίνεται να προτείνουν ορισμένοι, τότε χάνει αυτά τα χαρακτηριστικά και τη λογική ύπαρξή του. Και γι' αυτό και η πρόταση της Κομισιόν ήταν να διατηρηθεί το status quo όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής. Και δεν θα θέλαμε Είμαστε απρόθυμοι να διευρυνθεί στη στέγαση ή στην απόδοση της ενεργειακή αποδοτικότητα. Όχι γιατί δεν θα θέλαμε να αναπτυχθούν αυτοί οι τομείς, αλλά είναι τομείς που θα μπορούσαν να καλυφθούν κάλλιστα από το ΕΤΠΑ. για το θέμα της σύνδεσης με το CEF, τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Έχω σημειώσει τα σημαντικά σχόλια του εισηγητή για το ότι χρειάζεται να βρεθεί η σωστή βάση για το συγκεκριμένο θέμα. Φυσικά η Κομισιόν είναι ανοιχτή για να εξετάσει οποιαδήποτε διατύπωση συμβιβαστική που θα εξασφάλιζε ότι η διευκόλυνση αυτή θα έχει την υποστήριξη που χρειάζεται ώστε να δει το φως της ημέρας, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούμε μήπως υπάρξει απώλεια κάποιων από τα στοιχεία κλειδιά ε, κλειδιών μάλλον της ε, διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη που θα φύγουν στις εθνικές ε, χορηγήσεις γιατί όντως αφήνει περιθώριο για συγκεκριμένες προτεραιότητες. Αυτό είναι και άλλο στόχος, ότι μπορούμε δηλαδή να στοχεύσουμε που υπάρχει μια συγκεκριμένη ανάγκη για κάποια υποδομή. Και έτσι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε λοιπόν για έναν μηχανισμό που θα σήμαινε την απώλεια αυτής της δυνατότητας. Τώρα, για το συγκεκριμένο δημοσιονομικό θέμα, εδώ βεβαίω θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τελική δομή του προπολογισμού, Αλλά η ε, δική μου αντίδραση θα ήταν ε, ότι αν εντάξουμε μέσα στο τελικό πουδοπό και τη σχετική νομοθεσία τη συγκεκριμένη διάταξη για τη χρήση της διευκόλυνσης ιδιώντας την Ευρώπη στον τίτλο 1α για 10 δις ή οποιοδήποτε άλλο αριθμό από το, το, Ταμείο Συνοχής που προέρχονται από το 1β είναι δυνατόν. Αν ο νομοθέτης αυτό αποφασίζει τότε αυτό αποτελεί την βάση για την υλοποίησή του. Από τη στιγμή που θα μεταφερθεί λοιπόν στο η διευκόλυνση τότε πια δεν θα είναι χρήματα του Ταμείου Συνοχής, χάνουν τα χαρακτηριστικά του Ταμείου Συνοχής από τη στιγμή που μεταφέρονται. Εκτός από το γεγονός ότι κάποια ή μάλλον ότι οι κανόνε που ισχύουν για το Ταμείο Συνοχή θα εξακολουθήσουν να ισχύουν όσον αφορά δηλαδή τα ποσοστά χρηματοδότηση, στη χρήση και ούτω καθεξής. Ε, ε, αλλά εμπίπτει σε άμεση διαχείριση. Εφευρίσκουμε κάτι νέο εδώ, αλλά εμπίπτει στην άμεση διαχείριση και δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι χρήματα συνοχής υπό την άμεση διαχείριση. Είναι υπό το CEF, τη Διευκόλυνση Συνέντευξη στην Ευρώπη, γιατί διατηρεί κάποια χαρακτηριστικά της χρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής και αυτά είναι που οδήγησαν στην μεταφορά του κονδυλίου Τώρα, για τα όσα είπαμε εδώ ε, τώρα, είναι το θέμα είναι ότι, κοινή, ε, ότι ο ισχύοντας γενικός κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για όλα τα ταμεία ε, με τον ίδιο τρόπο. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στις περιφέρειες εδώ θα πρέπει να ισχύουν οι γενικές διατάξεις η σύνδεση με τα μακροοικονομικά στοιχεία που ορίζονται εδώ, εντάξει, εντάξει, καλά τα επιχειρήματα, αλλά εμείς δεν, θα στηρίζαμε μια τροπολογία που θα τα επανέφερε όλα αυτά απλώς στο Ταμείο Συνοχής. Έχουμε απομακρυνθεί από όλα αυτά πια και οι οικονομικές περιστάσεις τις οποίες όλοι γνωρίζουμε αιτιολογούν την προσέγγιση που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Κομισιόν. Το θέμα τώρα των κοινών δικτών Είναι καλύτερο να έχουμε κοινού δείκτες και να τους έχουμε σε όλα τα ταμεία σε εφαρμοστικές πράξεις, διότι έτσι είναι καλύτερος τρόπος για να έχουμε κοινού δείκτες. Ευχαριστούμε. Ο Βίκτορ. it's okay. Good. On uh, the comments... Θέλω πρώτα απ' όλα να πω στην κυρία Ματσόνη, έφυγε βέβαια, αλλά φυσικά και είμαι υπέρ του να προχωρήσουμε προς μια οικονομία βασισμένη σε χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Αυτό είναι ο προσανατολισμός, η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και εκπομπών ε, του θερμοκηπίου. Είναι και δικιά μου δέσμευση αυτή. Και γι' αυτό και είμαι διατεθειμένος να δουλέψω προς αυτή την κατεύθυνση ενσωματώνοντας τις τροπολογίες της. Όσον αφορά τώρα όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές μεταφορών. Και πάλι έχω την τάση να επικεντρωθώ στα, στις κύριες υποδομές των ε, ευρωπαϊκών δικτύων. Να μην δουλέψω δηλαδή με δίκτυα τα οποία έχουν να κάνουν με τις περιφέρειες ή με τμήμα των περιφερειών. Όσον αφορά τα σχόλια του Έλληνα συναδέρφου του κ. Χρυσόγελου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια. Όπως ξέρετε πολύ καλά, εγώ ίδιος έχω υποβάλει τροπολογίες προκειμένου να ενισχύσω την προστασία της βιοπικιλότητας και του Natura 2000. Έκανα επίσης ό,τι μπορούσα προκειμένου να αναφέρω ξανά και ξανά την βελτίωση της διοικητικής και θεσμικής ικανότητας. Είμαι έτοιμος να δω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, να είναι και εκείνη έτοιμη με ένα εφικτό, αποτελεσματικό σχέδιο και αυτό να το κάνει πριν από το 2014. Γιατί θεωρητικά αυτό σημαίνει ότι η θεσμική και διοικητική ικανότητα το 2014 πρέπει να είναι ήδη έτοιμη και να λειτουργεί. Και όπως ακούσαμε και σήμερα εδώ σε αυτή την αίθουσα, εμείς οι ευρωβουλευτές μερικές φορές χρειαζόμαστε επεξηγήσεις για το τι ακριβώς σημαίνει μία έννοια ή μία πρόταση. Αν πρέπει να έχουμε εδώ πέρα την Βρυτάνικα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια εγκυκλοπαίδεια δηλαδή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταλαβαίνετε τι θα χρειαστούν τότε στις περιφέρειές μας. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τη θεσμική και τη διοικητική ικανότητα και να το κάνουμε τώρα. Γιατί αυτό είναι γενικότερο. Όσον αφορά τώρα τις μεταφορές που είπε ο κύριος Χρυσόγελος και πάλι να ξέρετε ότι εγώ είμαι έτοιμος να συνεργαστώ, αλλά μην ανοίξουμε υπερβολικά την ψαλίδα, να επικεντρωθούμε σε ότι είναι διευρωπαϊκό, όχι σε άλλες πτυχές. Θα βρω έναν τρόπο πάντως να συντάξω μια συμβιβαστική πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα πώς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις κλιματικές αλλαγές. Ε, εγώ χαίρομαι που ένας από τους συναδέλφους από άλλη πολιτική ομάδα δήλωσε ότι είναι κάποιο είδους πράσινη επανάσταση αυτή η έκθεση για το Ταμείο Συνοχής. Πολύ χαίρομαι, γιατί πράγματι αντικατοπτρίζει αυτό το πνεύμα όλων των πολιτικών ομάδων. Επιτέλους πρόκειται για μια ευρωπαϊκή αξία, πραγματική ευρωπαϊκή αξία. Γι' αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να το βάλουμε εδώ και στο Ταμείο Συνοχής. Για τα υπόλοιπα, για τα σχόλια του κ. Ολμπρίχτ. Φυσικά και θέλω να επικεντρώσω το Ταμείο Συνοχής σε αυτό για το οποίο προορίστηκε από την αρχή. Και η δικιά μου ιδέα να ανοίξουμε στην επιλεξιμότητα ε, προγράμματα που έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργειας των νοικοκυριών, τη θέρμανση και ε, εργοστάσια, προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το κάνω για δύο λόγους. Και το λέω αυτό και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν το είχαμε κάνει αυτό μέχρι σήμερα, ίσως να έχει λυθεί το πρόβλημα. Αλλά αν κοιτάξουμε τις στατιστικές που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μας λένε ξανά και ξανά ότι με τις τρέχουσες ε, επενδύσεις, με την τρέχουσα χρηματοδότηση και με τους τρέχοντες κανόνες επιλεξιμότητας φτάνουμε στο 2020. Άρα στο τέλος της επόμενης δημοσιονομικής ε, περίοδου μόνο ο μισός προϋπολογισμός θα έχει βελτιώσει την εξοικονόμηση ενέργειας, ε, θα έχουν μειωθεί στο ίμιση e οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κλπ. κλπ. Είναι ζωτική σημασία λοιπόν να δώσουμε όθηση στο πρασίνισμα όχι μόνο της οικονομίας μας, αλλά να ετοιμάσουμε την οικονομία μας ώστε να είναι βιώσιμη. Και γι' αυτό και πρότεινα τις τροπολογίες μου που αναφέρονται στην εξοικονόμηση ενέργειας από τα νοικοκυριά, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα επιλεξιμότητας και για τα ε, δίκτυα μεταφορών θέρμανσης και για να απαντήσω και στον κύριο Χρυσόγελο επ' αυτού, όλα τα σχέδια τα οποία βασίζονται στις ανανόσιμες πηγές ενέργειας είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τις τροπολογίες μου. Και δεν πειράζουμε εδώ πέρα καθόλου το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Είναι απόλυτα επιλέξιμες οι ανανόσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να είναι εκτός από τον ηλεκτρισμό. Δεν θέλουμε δηλαδή να πειράξουμε καθόλου το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Έτσι, έχουμε σταθερότητα για ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί. Την καύση δεν τη συμπεριλαμβάνουμε. Τώρα, άλλες πτυχές. Για το CF. Συμφωνώ με τον κύριο Όλμπριχτ και δεν είναι τυχαίο. Τα προβλήματά μας που αναφέρθηκαν και από την κυρία Ματσόνη, τι είναι, λένε ότι έχουμε ένα πρόβλημα και μπορούμε να έχουμε τώρα συμβιβασμό. Πρέπει να πετύχουμε συμβασμό για τη χρηματοδοτική διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Αν δεν υπάρξει συμβιβασμός, τότε το σχέδιο αυτό πάει πέθανε. Και εγώ δεν θέλω η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη να έχει αυτή την τύχη. Εγώ θέλω να δώσει καρπούς αυτό για το οποίο αρχικά ε, προβλέπεται για την ε, διασυνοριακή αυτή διάσταση. Είναι πολύ σημαντικό. Κάνω έκκληση λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επίτροπη να πετύχει τον συμβιβασμό αυτό που θα στηρίξουμε και πιστεύω και το Συμβούλιο. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και εδώ το Συμβούλιο είναι πολύ πιο κοντά στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από ό,τι Κομισιόν. Υπάρχει τεράστια ανάγκη να πετύχουμε τον συμβιβασμό αυτό. Τέλος, για τα 10 δισεκατομμύρια που αναφέρθηκαν από τον κύριο Βλάσακ, τον οποίο και θέλω να ευχαριστήσω για τα θετικά του σχόλια. Μα είναι προφανές. Τα χρήματα πρέπει να βγουν από το Ταμείο Συνοχής. πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι της συνοχής θα τηρηθούν ακόμα και όταν μεταφέρουμε τα χρήματα στο συνδέοντα στην Ευρώπη. Και αυτή είναι η εκκλησία μου, γι' αυτό και ζητάω συμβιβασμό. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε καλούς συμβιβασμούς στο τέλος και ότι θα ψηφίσουμε την έκθεση με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου αυτό χρειάζεται ή με το Συμβουλίο όπου αυτό χρειάζεται. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και είμαι ανοιχτός για να ετοιμάσουμε μαζί τους συμβιβασμούς. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη που εδώ έχουμε τις λιγότερες τροπολογίες. Ο Ακίμ, ελπίζω να μην έχουμε μείνει δυο μας στην αίθουσα για να ακούσουμε την έκθεση αυτή, ότι θα παραμείνουν στην αίθουσα και οι συνάδελφοι. το λόγο. Όντως, Πρόεδρε, πέρα από τις τροπολογίε που έχω υποβάλει εγώ, μόνο 28 επιπλέον έχουμε. Σκέφτηκα ότι αυτό απεδείκνει πως είχαμε ήδη ε, συζητήσει αρκετά από μακρόν αυτή τη συζήτηση εδώ. Είχαμε οργανώσει και ακρόαση για το θέμα και ε, ε, είδαμε ότι η Επιτροπή ήδη έχει λάβει υπόψη τις <clears throat> απόψεις μας. Και φαίνεται να είναι όλοι πάνω κάτω ικανοποιημένοι. Όσον αφορά τις τροποποιήσεις των συναδέλφων, θεωρώ ότι κάποιες αλλαγές, θα μπορούν, βελτιώσεις θα μπορούσαν ακόμα να γίνουν. Ζητάμε, ας πούμε, να λαμβάνονται υπόψη το, να λαμβάνονται υπόψη οι ΟΕΣ σε περίπτωση διαγωνισμών γιατί θα πρέπει να σταματήσουν ε, οι διακρίσεις κατά των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας. Οι ε, ΕΟΕΣ είναι οργανισμοί που συμπεριλαμβάνουν ήδη εταιρείε από πολλές χώρες και θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Έπειτα υπάρχουν κράτη-μέλη, περιφέρειες όπου οι υπηρεσίες της Κομισιόν χρησιμοποιούν περισσότερο τους ΕΟΕΣ και θα πρέπει να γνωρίζουν καλύτερα ποιο είναι αυτό το μέσο. Έχουμε επίσης άλλα μέσα όπως το μέσο ε, Ευρωπαϊκής Εταιρικής Συνεργασίας ή το μέσο ένταξης που αφορούν βέβαια και τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Εγώ υποστηρίζω και μία μεγαλύτερη στόχευση σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος σε παραμεθόριες περιοχές όπου εκεί πρέπει και, θα, και μπορούν να αναπτυχθούν σημαντικά. Και μεγαλύτερη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και σε υφιστάμενα προγράμματα και σε μελλοντικά. Βέβαια, η κοινωνία των πολιτών είναι ένας αόριστος όρος και κάποια διευκρίνηση θα χρειαστεί. Με βέβαια κάποιο άνοιγμα σε οργανώσεις διαφόρων ειδών που θα πρέπει να ξεπερνά και τα όρια Τον... Ε, το ίδιο, τα ίδια ισχύουν βεβαίως και για τον σχεδιασμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τώρα, δεν μπορώ να συμφωνήσω με ορισμένε τροπολογίε των συναδέλφων. Η πρόταση τη Κομισιόν αλλά και το σχέδιο εκθέσεως δεν προβλέπουν να δοθούν περαιτέρω οικονομικά ε, κίνητρα για την ίδρυση και άλλων ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας. Αρκούν τα κίνητρα που υφίστανται για την ώρα, έτσι θεωρούμε, και νομίζω ότι δεν μπορώ να λάβω υπόψη μου το αίτημα αυτό. Τώρα είναι κατανοητή βέβαια η επιθυμία για την βελτίωση της διοίκησης του προσωπικού. Εκεί προβλέπεται και κάποια ευκαμψία. Τα δε αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλουν να εφαρμοστούν με παρόμοιο καταστατικό του προσωπικού όπως των ευρωπαϊκών οργανισμών έχει ωστόσο, ενέχει ωστόσο τον κίνδυνο ότι θα έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα λόγω του υψηλού κόστους ε, αποτρεπτικό χαρακτήρα για την ίδρυση και άλλων ΕΟΕΣ, Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας. Θεωρώ επίσης ότι η προθεσμία των έξι μηνών που προτείνεται στον κανονισμό είναι ισορροπημένη και μπορεί να επιτευχθεί με συμφωνία του Συμβουλίου ούτε παράταση, ούτε, ε, επιβράχη, ε, ούτε, ούτε ε, μείωση της προθεσμίας αυτής θεωρώ ότι είναι κατάλληλη, ότι είναι ορθή. Βέβαια, θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις υπερπεριφερειακές περιοχές και να χρησιμοποιήσουν και αυτές ενδεχομένως τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους εταιρικής Συνεργασίας για ε, την λειτουργία τους. Και αυτές οι outermost regions μπορούν ήδη να ιδρύσουν ΕΟΕΣ και ε, διαπεριφερειακά. Η στόχευση και ο καθορισμός ειδικών στόχων, αυτό, απέναντι σε αυτό τάσσομαι, ε, στέκομαι κριτικά. Διότι ναι μεν επιτυγχάνονται κάποιες πρόοδοι με τους ΕΟΕΣ, αλλά το εργαλείο αυτό είναι πολύ ανοιχτό και δικαίω είναι διαμορφωμένο πολύ ανοιχτά δηλαδή για να μπορεί να λάβει υπόψη και μελλοντικέ προοπτικέ, μελλοντικέ εξελίξεις. Αυτή η ευκαμψία και ο ανοιχτό χαρακτήρα πρέπει να διατηρηθούν. Ευχαριστώ λοιπόν όλε και όλου που κατέθεσαν τροπολογίε και αναμένω την περαιτέρω συζήτηση. και μια επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Και μετά βεβαίως αναμένω με ενδιαφέρον την αντιπαράθεση με το Συμβούλιο που σίγουρα θα ε, γίνει μάλλον πιο περίπλοκη από τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν εδώ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Είναι να δώσω το λόγο στους βοηθούς, αλλά κανείς δεν θέλει να, δώσει, να πάρει το λόγο. Εντάξει, το καταλάβαμε, τώρα η Κομισιόν. Α, όχι, πρώτα ο Γιάνν Όλμπριχτ, συγγνώμη. Είμαι σε πολύ ιδιαίτερη θέση γιατί ήμουν εισηγητής για τους ε, ομίλους αυτούς πριν από κάποια χρόνια και ξέρω πόσο δύσκολη ήταν η έγκρισή τους στο Συμβούλιο. Γι' αυτό και τα όσα κάνει ο συνάδελφος Τσέλερ είναι πολύ καλό βήμα μπροστά. σε σχέση με το ρόλο των ΕΟΕΣ και κατά πόσο θα είναι, πρέπει να είναι στο πακέτο της συνοχής ε, ή όχι. Γιατί δεν είναι τα χρήματα, είναι ένα νομικό μέσο. Εγώ νομίζω θα πρέπει να μπει στο πακέτο. Και η τροπολογία που πρότεινε ο Γιωακίμ Τσέλερ, είναι σημαντική γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε το πιθανό ρόλο των ΕΟΕΣ πέρα από το ρόλο της ολοκλήρωσης. Αυτό το μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους λόγους και όχι μόνο για διασυνοριακά που ήταν η αρχικός στόχος. Ως νομικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί λοιπόν για διάφορους λόγους, για διάφορους σκοπούς, αλλά δεν συμφωνώ με κάποιες από τις τροπολογίες που λένε ότι η οι ε, υπάλληλοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όσο πως και οι υπάλληλοι της Ένωσης. Περιμένω εδώ να δω την αντίδραση του Συμβουλίου. που σίγουρα θα είναι αντίθετο για μισθούς όπως τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς έως ας πούμε για ανάμεσα στην Πολωνία και τις Σλοβακίες με μισθούς ε, των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών θα ήταν πολύ εντυπωσιακό αν γινόταν όντως. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα για το πώς ε, θα εισαχθεί ένα ευρωπαϊκός θεσμός με, νομική, με νομικό πρόσωπο με διάφορες μεθόδους. Αυτό που είναι σημαντικό και η πρόταση του king Ζέλερ προέρχεται και από τις επαφές με την ε, αρμόδιους ε, για τη συνοχή που έχουν και τη λειτουργία της παρακολούθησης του ΕΟΕΣ. Παρακολουθούν, έχουν τις εκθέσεις, έχουν τα στοιχεία και βεβαίως το θέμα είναι τώρα τι πρέπει να αλλάξει. Και τώρα νομίζω αν καταφέρουμε στο Κοινοβούλιο να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο για να ενισχυθούν κάπως οι ΟΕΣ θα είναι μεγάλη επιτυχία γιατί η δισταγμή για αυτό το μέσο ήταν πολύ μεγάλη. Αλλά νομίζω πως προχωράει καλά. Βεβαίως, για το Συμβούλιο, το καλύτερο θα ήταν πέντε χρόνια. Όσο γίνεται δηλαδή περισσότερο. Αλλά για μας θα πρέπει να είναι λογικό, ας πούμε έξι μήνες. Ξέρω ότι προτάθηκε τέσσερις μήνες μόνο, αλλά δεν νομίζω πως το Συμβούλιο θα συμφωνήσει. Αν καταφέρουμε να έχουμε έξι μήνες, θα είναι ήδη μεγάλη επιτυχία. Ο κανονισμός λοιπόν αυτό δεν αφορά χρήματα, αφορά τη δημιουργία νέων πολύ ενδιαφέροντων μέσων με πολύ ευρύτερε λειτουργίες για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε κατάλαβα, ο David Sweet ε, έφτασε, κατέφτασε. Εκείνο γνωρίζει τα θέματα αυτά και μπορεί να πάρει και το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένα και δεν άκουσα. Ε, κοιτάξτε, εμεί ε, τελειώσαμε πολύ γρήγορα. Είστε πολύ, πολύ αποτελεσματικοί, όπω συνήθω. Ε, Κοιτάξτε, ε, δεν θέλω να πω και πολλά γιατί το μήνυμά μου δεν είναι διαφορετικό από τα όσα ήδη είπατε στην Επιτροπή σας. Ε, όπως ε, συνήθως εκτιμάμε τη θετική ανταπόκριση από, τους, από τον εισηγητή και τους υπολείπους που πήραν το λόγο στην Επιτροπή. Καταλαβαίνουμε ότι υποστηρίζει τόσο την αρχή όσον αφορά αυτό το μέσο και τους στόχους των αλλαγών μας και είμαστε γνώμονες γι' αυτό. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες τροπολογίες που ήταν υπό συζήτηση σήμερα, πολλές από αυτές γίνονται μέσα στο πνεύμα γίνονται μάλλον με καλή πρόθεση, αλλά σε ορισμένε περιπτώσει έχουμε επιφυλάξει. Γιατί η σύνταξη τη ε, τροπολογία εκφράζει μια πολιτική βούληση, αλλά χωρί να το τοποθετεί με συγκεκριμένα, να λέει μάλλον με συγκεκριμένα λόγια τι θα σημαίνει αυτό στην εφαρμογή του κανονισμού. Δηλαδή, είναι μια αναφορά σε μια τηλογική σκέψη, για παράδειγμα, που δεν έχει όμω πρακτικό αντίκτυπο. Ίσως αυτό να είναι βοηθητικό από πολιτικής άποψης, αλλά όχι απαραίτητο για την εφαρμογή του κανονισμού. Μια δεύτερη ομάδα τροπολογιών αφορά τροπολογίες που φαίνεται να εστιάζονται σε, μια συγκεκριμένη πτυχή όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι ΕΟΕΣ. Και εδώ θα ήθελα να θυμίσω στην Επιτροπή ότι στον τροποποιητικό κανονισμό στόχος μας είναι να καταστεί ευκολότερη χρήση των ΕΟΕΣ και να είναι και πιο εύκαμπτη Γι' αυτό και δεν θέλουμε να εγκρίνουμε τροπολογίες που φαίνεται να τονίζουν ή να ευνοούν ε, μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο είδος ομαδοποίησης ε, ακόμα και αν είναι θετικός ο τρόπος ομαδοποίησης, δεν χρειάζεται να αναφέρεται ξεχωριστά. Έπειτα, ο αντίκτυπος ε, του κανονισμού ΕΟΕΣ στον δημοσιονομικό κανονισμό Μπορεί να είναι ο ορισμό ή μπορεί να αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως στην έρευνα, στην περιβάλλον ή αλλού. Και θα ήθελα να θυμίσω στους κύριους βουλευτέ πως αυτός ο κανονισμός αφορά το λειτουργία του μέσου ΕΟΕΣ και δεν μπορεί να αλλάξει ο ίδιος τους κανόνες άλλων ευρωπαϊκών κανονισμών. Στόχο, ωστόσο των συγκεκριμένων τροπολογιών ήδη είναι προσαρμοσμένος και ήδη είμαστε σε επαφή με του διαχειριστές των άλλων πολιτικών και βλέπουμε οποιαδήποτε εμπόδια ε, και φροντίζουμε μάλλον ώστε να αρθούν οποιαδήποτε εμπόδια. Τέλος υπάρχουν τροπολογίες που είναι οι καλές τροπολογίες που θα έλεγα είναι απόλυτα αποδεκτές και θα ακολουθούν την κατεύθυνση που θέλουμε. Ίσως εμείς για λόγους της Επιτροπής να μην αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τόσο πολύ, αλλά αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη στηρίξει, ίσως ε, και να καταστήσουν το κείμενο μας ακόμα πιο σαφές. Γι' αυτές είμαστε ευχαριστημένοι. Τώρα, αν το Συμβούλιο των Υπουργών θα τις δεχτεί, ε, θα δούμε. Αυτά είναι συντομία κυρία Πρόεδρε, η θέση μας για αυτές τις τροπολογίες. Αν έχετε ερωτήσεις ή αν θέλετε να τις συζητήσουμε, ο συνάδελφος που μόλις έφτασε και εκείνος και είναι πιο αρμόδιος για να μιλήσει για συγκεκριμένα ε, θέματα, είναι παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τις επισημάνσεις του Γιάνν Όλμπριχτ που όπως και η πρόεδρός μας τότε ως επίτροπος ήταν ας πούμε μέες του συστήματος. Τώρα βέβαια έχει ξεφύγει από το επίπεδο του βρέφους, από την ε, βρεφική ηλικία το σύστημα. Υπάρχουν 26 ε, μονάδες που λειτουργούν και ε, από την Τσεχία και με την Αυστρία και ο EOS είναι βέβαια ένας τρόπος να εμβαθύνει αυτή η συνεργασία. Βλέπουμε δηλαδή ότι η σκέψη να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες προσφέρει αυτό το νομικό εργαλείο, αυτή η σκέψη αναπτύσσεται και καταλαμβάνει όλο και περισσότερους, ε, περισσότερο χώρο ας πούμε. Πάντως ειδικά για τη Γερμανία βλέπω ιδιαίτερα στα ομοσπονδιακά κρατήδια να υπάρχει ο φόβος ότι κάτι τι θα χρειαστεί να δώσουν και γι' αυτό οι αντιστάσει είναι μεγαλύτερε. Να καταστήσουμε σαφέ στου υπεύθυνου εκεί ότι δεν πρόκειται να του πάρουν τίποτα, δεν πρόκειται να δώσουν τίποτα. Πρόκειται απλά για μια βελτίωση τη διαμεθοριακής συνεργασία. Αν πετύχουμε να το κάνουμε σαφέ αυτό, τότε νομίζω ότι ο ΕΟΕΣ θα αποδειχθεί στο μέλλον το πιο σημαντικό εργαλείο για την διαμεθοριακή συνεργασία. Και έτσι θα έχουμε βάλει ένα ακόμα ορόσημο προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Επ' αυτού, με ναι, αυτό μάλλον, κλείνουμε και αυτό το θέμα. Πρόκειται για την τελευταία μας ε, συνεδρίαση και συζήτηση πριν από τη μεγάλη ψηφοφορία ε, του Ιουλίου. Ε, δεν ξέρω αν ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μας δώσει τις ευλογίες της στην παραπέρα αυτή πορεία. Κυρία Πρόεδρε, θα επαναλάβω ίσως τα όσα είπα χθε ότι η Κομισιόν είναι στη διάθεσή σας για τις επόμενες ημέρες και βέβαια στην διάθεση του εισηγητή για τους διάφορους κανονισμούς, αν χρειαστεί δηλαδή από άποψη τεχνική να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο στα πλαίσια της διαδικασίας που θεωρούμε ότι θα είναι βέβαια δύσκολη, θα χρειαστεί να εξετάσουμε όλες τις τροπολογίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη επιθυμείτε για βελτίωση της κατανόησης, είμαστε στη διάθεσή σας. Είδα από τις χρησινές και σημερινές ε, συζητήσεις ότι οι τροπολογίες κατατίθενται. Βλέπω και με ποιο τρόπο τις εξετάζει ο εισηγητής. Αυτά μας καθησυχάζουν σχετικά με το τι θα προκύψει από την ψηφοφορία του Ιουλίου για την περαιτέρω συνεργασία των θεσμικών οργάνων. Βλέπουμε δηλαδή να είναι να υπάρχει κατανόηση για τα διάφορα θέματα που προκύπτουν και νομίζω ότι θα μπορέσουμε με συνεργασία να βρούμε μια ικανοποιητική λύση. Δεν βλέπουμε δηλαδή για ποιο λόγο άραγε να μην είναι δυνατόν να βγούμε από τη διαδικασία αυτή με ένα ξεκάθαρο σύνολο κανόνων που να εξυπηρετεί την άσκηση της πολιτικής αυτής. Βρίσκω ότι έχουμε μια κοινή ενατένιση των κοινών αυτών στόχων. Γι' αυτό και σας υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ Νικόλαε θα περάσουμε το μήνυμα και στους άλλους εισηγητές ώστε να μπορέσουν να υποφεληθούν από την τεχνική σας υποστήριξη. Εδώ λίγη η συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 11 και 12 και τι όμορφα που είναι να είναι μικρή η Επιτροπή. Δουλεύουμε πολύ καλύτερα και γρηγορότερα όταν είμαστε λιγότεροι. Να το κάνουμε λοιπόν τη συνεδρίαση μας πάντοτε Πέμπτη ή Παρασκευή απόγευμα. Ευχαριστώ όλες και όλους. Διακόπτη τη συνεδρίαση.